Ladies and gentlemen, dear colleagues, have a seat, please. Nous avons droit à une... Αγαπητοί συναδελφοί, καθίστε παρακαλώ. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αίθουσα που αντιστοιχεί στο κύρος και στη σημασία της Επιτροπής Προπολογισμών, που όμως ε, για την ώρα δεν αντιστοιχεί στον αριθμό των παρόντων μελών και στην σημασία του ακροατηρίου. Γι' αυτό σας παρακαλώ να καθίσετε όσο γίνεται πιο σύντομα και να θυμίσω στους ακροατές ότι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι θα πρέπει να παραμείνουν σιωπηλοί. Έχουμε δύο μισές ημέρες συνεδρίασης. Πριν να αρχίσουμε την εξέταση της σημερινή διάταξη, ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στον συνάδελφο Γιάσεκ Βλόζοβιτς, δεν ξέρω αν είναι ήδη εδώ, αλλά χθε είχε τα γενέθλιά του. Μπορείτε κι εσείς να του ευχηθείτε. Εγώ το εύχομαι στο όνομα όλης της Επιτροπής. Χαιρετίζω την παρουσία του Γενικού Διευθυντή Προπολογισμού μας κάνει την τιμή να είναι παρόν σήμερα. Μου είπε ότι δεν θα μπορεί να είναι εδώ αύριο το πρωί γιατί συνεδριάζει το σύνολο των επιτρόπων και γι' αυτό και εκτιμούμε την παρουσία του εδώ απόψε. Είδατε το σχέδιο μερικής διάταξης, κάποιες μικροαλλαγές θα πρέπει να γίνουν. Λάβατε ένα φάκελο και επίση ένα συμπληρωματικό φάκελο με μεταξύ άλλων ένα σημείωμα σε σχέση με την βοήθεια προς την ΑΕΤ μετά από την τραγωδία του σεισμού. Θα εξετάσουμε αυτό το σημείο στο σημείο 19 της ημερήσιας διάταξής μας αύριο το πρωί τη παρουσία εκπροσώπων της Επιτροπής. Ο κύριος Μαντζερβίζη που είναι Γενικός Διευθυντής για την Ανάπτυξη και ο κύριος Τσάγγελ που είναι Γενικός Διευθυντής της ΕΚΟ. Και φυσικά κάλεσα τους συναδέλφους από τις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και από την Επιτροπή Ανάπτυξης ώστε να παρακολουθήσουν, να συμμετέχουν. Να στείλουν τουλάχιστον κάποιον εκπρόσωπο της επιτροπή του, ώστε να παρακολουθήσουν αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμβάλλει στην ανακούφιση του πληθυσμού που χτυπήθηκε από αυτή τη θεομηνία. Κάποιες επίγουσες προβλέψεις ήδη έχουν γίνει από την Κομισιόν ή μπορεί να γίνουν, αλλά από τη στιγμή που θα υπάρχει η κατάλληλη χρηματοδότηση. Χρειάζεται η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχουν επίγουσες διαδικασίες ε, που μπορούμε να ακολουθήσουμε και θα δούμε που βρισκόμαστε αύριο το πρωί. Στο 19, όπως είπαμε, τις μερίσεις διάταξης. Για απόψε, μια μικρή αλλαγή μετά από έτοιμα του εισηγητή, το σημείο 7, για τον υπολογισμό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, συγητής είναι ο κύριος Ζαν Λικντε Άννα, Θα εξεταστεί λοιπόν μετά από το σημείο 8 και 10. Το ίδιο, σημείο, ε, ε, το ίδιο συμβαίνει και για το 9. Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Και το σημείο 11 για το ΣΥΣ, Σένγεν 1 δεύτερη γενεά, θα αναβληθεί για μια άλλη συνεδρίαση μετά από αίτημα του εισηγητή του κ. Άλβαρο που χρειάζεται κάποιο παραπάνω χρόνο. Από το πρωί θυμίζω ότι σύμφωνα με την παράδοση της Επιτροπής μας θα ξεκινήσουμε το πρωινό, το δεύτερο μισό δηλαδή της συνεδρίασής μας με ψηφοφορία. Οι ψηφοφορίε δεν υπάρχουν πολλές, τρει προβλέπονται και είναι πιθανόν να γίνουν μόνο δύο. Θα πρέπει να το δούμε σε λίγο στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών, την παρουσία του κυρίου Μάνκα που είναι ο εισηγητή για τον προπολογισμό του 2010 για να δούμε αν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε αύριο το πρωί δεδομένων των στοιχείων που λάβαμε πρόσφατα και που πιστεύουμε ότι χρειάζονται κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις πριν να είμαστε βέβαιοι ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα μπορέσει να ψηφίσει. Θα το δούμε στους συντονιστές λοιπόν και ο κύριος Μάνκα θα μας πει και εκείνος την άποψή του. Για το σημείο 14 και 13 θα ψηφίσουμε αύριο. Για το σημείο η κυρία Ναντέζντα Νέισκι δεν θα μπορεί να είναι μαζί μας όσον αφορά τις εξωτερικές υποθέσεις γιατί είχε ένα μικρό ατύχημα υγείας και από ό,τι κατάλαβα ο συνάδελφος Γκουαλτιέρη δέχτηκε να την αντικαταστήσει. Και όσον αφορά το σημείο 14 η Μόνικα Χολμάιερ είναι επίσης άρρωστη έχει πάθει κάποια είδος γρήπης που δεν είναι πολύ σοβαρή αλλά η συνάδελφος Γκρέσλε θα πάρει τη σκητάλη και θα μας θαμπώσει με τη συνείδητη της φράδια. Δεν έχουμε μεταφορές γιατί είμαστε στην αρχή του χρόνου και οι πιστώσεις βρίσκονται στις γραμμές που χρειάζονται δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, οπότε θεωρούμε πως ε, κλείσαμε το σημείο 1, εγκρίνουμε λοιπόν την ημερησία διάταξη, ανακοινώσει του Προέδρου, έχετε έναν κατάλογο με τις διαθέσιμες γλώσσες. Έχουμε σήμερα δυνατότητα να ακούμε ρουμάνικα. Δεν ξέρω γιατί θα τα έχουμε αύριο, οπότε εκμεταλλευτείτε το ακούσετε όλοι οι Ρουμάνικα σήμερα. Μεταδίδεται η συνεδρίασή μας στο ίντερνετ και όπως βλέπετε και στο Κόμπου News. Έχει δημοσιευθεί ο προπολογισμό 2010 στο site Aeroplex και έχετε τις διευθύνσεις εδώ. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 16 Νοεμβρίου 2009. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Θεωρώ ότι εγκρίνεται τα πρακτικά το ίδιο και στο σημείο 4 για τη συνεδρίαση 1ης και 2 ης Δεκεμβρίου 2009. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 5. Ετήσια έκθεση 2008 για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας πρέπει να γνωμοδοτήσουμε ως ήθιστε και δίνω το λόγο στον κύριο Κουαλτιέρη. Παρακαλώ. Ε, Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως θυμήσατε, εγώ και η συνάδελφος Νέισκη ως μόνιμη εισηγητές για τον προπολογισμό της κοινή εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής Άμυνα. Ε, συνεργαστήκαμε ε, φέτος υπογράψει την έκθεση η κυρία Νέισκη και εγώ απλώς θα σας ενημερώσω. Καταρχήν έχουμε τα αριθμητικά στοιχεία. Το 2008 ήταν μια χρονιά ρεκόρ με την έννοια ότι ο προπολογισμό έφτασε στα 289 εκατομμύρια με σημαντική αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Φτάσαμε σε υψηλότερο επίπεδο ακόμα και από τους επόμενου ε, διαδοχικούς προπολογισμού. Ωστόσο, πρόκειται και αυτό για μια σειρά από λόγου. Ήταν ένα έτος διαφόρων ε, πολύ δεσμευτικών ε, αποστολών όπω το Κωσυφοπέδιο, το Αφγανιστάν, η Γεωργία και ωστόσο υπογραμμίζεται τόσο στην έκθεση του Αλμπερτίνη όσο και στη δική μας νομοδότηση, στο σχέδιο γνωμοδότησης, πως πρόκειται για έναν ε, νούμερο μικρό κάτω από το 4% του τίτλου 4 και νομίζω ότι θα μπορέσουμε αργότερα να υποβάλουμε μια τροπολογία σε σχέση με αυτή τη διατύπωση, να αναδιατυπώσουμε αυτή την πρώτη παράγραφο και να μην περιοριστούμε στο να υπογραμμίσουμε αυτό τον περιορισμένο προϋπολογισμό ΚΕΠΑ σε σχέση με τις πολύ μεγάλες υποχρεώσει που έχει να αντιμετωπίσει η Ένωση, αλλά και σε σχέση με τις ανησυχίες μας για αυτό το περιορισμένο, το, το μικρό μάλλον ε, κονδύλι. Δεύτερο σημείο στο σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Νεΐσκη αφορά την διοργανική συμφωνία όπου υπογραμμίζεται ο περίεργος χαρακτήρας ε, του προϋπολογισμού ΚΕΠΑ ε, μέσα στο πλαίσιο του, της Διοργανικής ε, Συμφωνίας, το σημείο 42, στο πλαίσιο μιας γενικότερης ανησυχίας που έχουμε για την αντίφαση ανάμεσα στον διακυβερνητικό χαρακτήρα σε σχέση με τις διαδικασίες απόφασης της ΚΕΠΑ και το γεγονός ότι χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των ε, δημοσιονομικών διαδικασιών. Τέλος, τα άλλα σημεία αφορούν ε, τις διαδικασίες διαβούλευσης που προβλέπονται περιοδικά από την Διοργανική Συμφωνία του 2006 ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις ε, ΚΟΠΣ. Εμείς θέλουμε να διευρύνουμε το χαρακτήρα αυτών των διαβουλεύσεων έτσι ώστε να είναι και πιο ακριβής ο προϋπολογισμός για τις αποστολές που ήδη έχουν ολοκληρωθεί και να έχουμε έτσι και τη δυνατότητα μιας ανάλυσης που θα μας επιτρέψει να συνδέσουμε την αξιολόγηση του κόστους των αποστολών PESC PESD με τον αντίκτυπο των άλλων ε, χρηματοπιστωτικών μέσων της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα υπάρχει και ένα κομμάτι της γνωμοδότησης που, που μιλά για τις πρωτοβουλίες για την βελτίωση του κόστους, ε, βελτιστοποίηση μάλλον του κόστους της ΚΕΠΑ και συνδέεται με το γεγονός ότι η απουσία κοινών διαδικασιών για την ε, κατάρτιση και για την ε, πρόσληψη προσωπικού στα κράτη-μέλη πολιτικού προσωπικού οδηγεί στην αύξηση του αριθμού του προσωπικού που βρίσκεται υπό άμεση σύμβαση της Ένωσης που φυσικά οδηγεί σε μεγαλύτερο κόστος για αυτό το προσωπικό. Έτσι λοιπόν ζητάμε την ανάπτυξη πρωτοβουλειών ώστε να διευκολύνουμε την πρόσληψη ανθρώπων ε, με συμβάσεις σε εθνικό επίπεδο όταν πρόκειται για αποστολές ΚΕΠΑ και επίσης ζητάμε να αναλυφθούν πρωτοβουλίες ώστε να ενισχυθούν οι κοινέ δυνατότητες ε, στο πεδίο της ΚΕΠΑ ιδιαίτερα στο επίπεδο των ε, αποθηκών. Κάτι γίνεται σχετικά με το ε, στην Βοσνία και για τα μέσα μεταφορών επίσης. Υπάρχει και ακόμα μια παράγραφο ε, στη γνωμοδότηση όσον αφορά το κοινοβουλευτικό έλεγχο των ορισμού των ειδικών εκπροσώπων. Είναι μια ιστορική διεκδίκηση του Κοινοβουλίου και τελευταίο σημείο αφορά ο προβληματισμό μας για την έλλειψη διαφάνειας και ενημέρωσης τις αποστολές με ενωτικό χαρακτήρα που όπως αναφέρει και η συνθήκη δεν, χρηματοδοτούνται, δεν προβλέπονται να χρηματοδοτούνται από τον ε, κοινοτικό προπολογισμό, αλλά ωστόσο και υπό το φως άλλων άρθρων που ε, αναφέρονται στη συνθήκη της Λισαβόνας και προβλέπουν ε, ενεργό έλεγχο του Κοινοβουλίου για το σύνολο της ΚΕΠΑ και ΚΠΑ. θα ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί ο ρόλος ο ελεκτικός του Κοινοβουλίου για το σύνολο των αποστολών και άρα και για την υπόθεση των στρατιωτικών αποστολών. Μια άλλη τροπολογία εδώ υπάρχει, πιο τεχνική υφής, που θα ήθελα να σας την παρουσιάσω. Ότι δηλαδή στο κείμενο όπως έχει διατυπωθεί υπάρχει μια μικρή οριστία σε σχέση με την μνήμα στο άρθρο 41 παράγραφος Δέλτα του Συνθήκης του Λισαβόνα γιατί στην πράξη αυτό το άρθρο αποτελείται από δύο κομμάτια, δύο τμήματα. Εδώ αναφερόμαστε στο τμήμα που αφορά τη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο που με τη σειρά του κάνει μνήμα για την επιταχυμένη χρηματοδότηση των πολιτικών αποστολών ενώ για το Startup Fund όπως αποκαλείται για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών αποστολών που βαραίνει τα κράτη-μέλη η συνθήκη δεν προβλέπει διαβούλευση με το Κοινοβούλιο αλλά εμείς ακριβώς μέσα στο πλαίσιο των προηγούμενων ε, προβληματισμών θεωρούμε ότι και για αυτή τη διάσταση θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή του Κοινοβουλίου αλλά εδώ δεν πρόκειται για μια πραγματική τροπολογία, αλλά για τεχνικής φύσης αναδιατύπωση. Αυτό είναι το περιεχόμενο του σχεδίου γνωμοδότησης. Και φυσικά περιμένουμε τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Merci, Σας ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφε. Ήταν σαφέστατη και πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση αυτή για το σχέδιο της γνωμοδότησης και για τις προτινόμενες τροπολογίες. Μήπως θα ήθελε κανείς το λόγο. Ουδής. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για γνωμοδότηση απλώς και μάλιστα για το 2008 υπάρχει κάποια διαφορά με την επικαιρότητα, ιδιαίτερα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και η επικαιρότητα είναι πολύ σημαντική γιατί έχουν αλλάξει πράγματα. Παρ' όλα αυτά η γνωμοδότηση έχει μια πολιτική βαρύτητα γιατί θα καταρτιστεί και θα συζητηθεί στην Ολομέλεια ενώ προετοιμάζουμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή την ε, θέση σε ισχύ της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης με βάση τη συνθήκη Λισαβόνας, καθώς και το αξίωμα του είπα εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική. Άρα, η γνωμοδότηση αυτή και η ψηφοφορία που θα γίνει σχετικά στην επόμενη Ολομέλεια ε, για την έκθεση της αρμόδιας κατουσία επιτροπής που είναι η Επιτροπή Εξωτερικών θα είναι ευκαιρία να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να προτείνει κάποιους τρόπους βελτίωσης ε, της κατάστασης για το μέλλον. Αν δεν θέλει κανείς το λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γουαλτιέρη, να υπενθυμίσω ότι Σήμερα λίγη η προθεσμία για τις τροπολογίες, σήμερα στις 7 το απόγευμα, αύριο στις 9 το πρωί θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης με τις τροπολογίες. Στη συνέχεια θα υποβληθεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που θα εγκρίνει την κατουσίαν έκθεση στις 23 Φεβρουαρίου προκειμένου να, περάσουν, να περάσει στην δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου. Ωραία. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, τον προϋπολογισμό του 2011. Για τα Συγγνώμη, λεπτός, όχι τα λοιπά τμήματα. Καταρχήν, το γενικό προϋπολογισμό και τα λοιπά τμήματα στη συνέχεια. Για το βασικό προϋπολογισμό, η συγκήτρια είναι η κυρία Συντόνια Λουσμπιέτα Γεντζογεύσκα, στην οποία δίνω το λόγο για την παρθενική της ομιλία ως Γενικής Συγγήτριας για τον προϋπολογισμό. Θα σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω αγγλικά και όχι πολωνικά, γιατί για τα δημοσιονομικά θέματα έχω μεγαλύτερη άνεση στα αγγλικά όλος παραδόξως και όχι στη μητρική μου γλώσσα. Προς το παρόν λοιπόν θα μιλήσω αγγλικά. Όντως αυτή είναι η παρθενική μου ομιλία στην Επιτροπή αυτή προπολογισμών, ειδικά ως γενική συγγήτρια ε, για τον δικό μου προϋπολογισμό, γιατί θα σας εκφέρω τις προσωπικές μου ιδέες για το τι προτείνω για τον προϋπολογισμό του 2011 και περιμένω με ανυπομονησία τις ε, παρατηρήσεις σας μετά από τα δικά μου σχόλια και τις ε, προτάσεις σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα. Καταρχήν, να αναφερθώ στο πρωτόλιο έγγραφο που εκπονήσαμε με τον Λάζλο Σουριάν, που έχει τη μορφή εγγράφου εργασίας και έχει μοιραστεί, αν δεν κάνω λάθος, σε όλους σας. Ευχαριστώ θερμά τη Γραμματεία που πρόλαβε να συντάξει και να μοιράσει αυτό το έγγραφο έγκαιρα. Δεν είναι φυσικά η οριστική του μορφή, αλλά περιλαμβάνει ήδη μερικά σημαντικά θέματα για την ετήσια δημοσιονομική διαδικασία, όπω διαμορφώνεται μετά τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ο προπολογισμό του 2011 και η σχετική διαδικασία θα είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί ε, είμαστε πρωτοπόροι, καπανεί σε νέο έδαφο και πρώτη φορά θα επεξεργαστούμε έναν ετήσιο προπολογισμό δυνάμει των νέων συνθήκων, των νέων διατάξεων τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Αυτό το σχέδιο ε, εγγράφου θα είναι μια σκιαγράφηση ουσιαστικά των αδρών γραμμών και θεμάτων όπως προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας και από την κοινή διακήρυξη. Ήδη κάποια ζητήματα τα πραγματεύτηκε η κυρία Γκρέλ ε, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και έτσι έχουμε και τα τρία στοιχεία. Την ερμηνεία της συνθήκης της Λισαβόνας, το έργο της προκατόχου μου στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και την ερμηνεία της κοινή διακήρυξης όπως προέκυψε πέρυσι. Έτσι έχουμε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα που καλό θα είναι να το έχουμε υπόψη για να προσανατολίσουμε το έργο μας και να έχουμε και ένα χρονικό ορίζοντα και υπάρχουν και κάποια διαδικαστικά ζητήματα που άπτονται του νέου μας πλαισίου. Το έγγραφο αυτό δεν είναι πολιτικό, δεν έχει πολιτική αξία πολιτικής διακήρυξης. Ουσιαστικά είναι ένα βοήθημα για την εργασία μας. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω για το σημείο 6 ημερήσιας διάταξης είναι ότι χρειάζομαι τα σχόλιά σας γιατί εγώ ήδη έχω κάποιες ιδέες για το περιεχόμενο του προϋπολογισμού του 2011 και ελπίζω να με υποστηρίξετε και να ενστερνιστείτε τις απόψεις μου για το περιεχόμενο αυτού του προπολογισμού. Ω βασικά θέματα για τον προπολογισμό μου για το 2011 θα ήθελα να περιλάβω κάποια ζητήματα για την νεολαία. Οι νέοι και ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της, διακι... της ε, κινητικότητας ε, και της αναζήτησης ε, εργασίας, ιδιαίτερα της πρώτης θέσης εργασίας, πολύ ενδιαφέρον θέμα για του νέου και στα πλαίσια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, αλλά θέμα και κινητικότητα σε θέματα παιδείας. Η κινητικότητα των φοιτητών, των μαθητών, των μαθητευομένων ή των ερευνητών. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει πολλά προγράμματα και θα ήθελα να τα εξετάσω και να δούμε ποια επιδέχονται βελτιώσεις σε αυτό το προϋπολογισμό του 2011. Um, είναι πολύ σημαντικό επίσης να θεωρήσουμε το, τη νεολαία και ως εποδό και ως σύνθημα και κλειδί και για άλλα ζητήματα, για την έρευνα ας πούμε, αλλά και για την καινοτομία. Θα έχει επεκτάσει λοιπόν το θέμα της νεολαίας και σε άλλους τομείς. Αλλά είναι συναφές και με το θέμα της κοινωνικής ένταξης. Αυτές φυσικά είναι κάποιες σύντομες ιδέες που μου ήρθαν στο μυαλό. Θα ήθελα να σας ενημερώσω και για τις προκλήσεις της νέας περίοδου, γιατί θα έχουμε τη νέα επιτροπή, οπότε θα έχουμε την ετήσια στρατηγική πολιτικών. Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα απαντήσει, ε, δεν θα αντιδράσει στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα έχει τον πρώτο λόγο. Οπότε θα ήθελα να με βοηθήσετε να διατυπώσουμε αυτή την πρώτη διακήρυξη, τον πρώτο λόγο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τη μορφή κατευθυντηρίων γραμμών για τον προπολογισμό. Και ελπίζω στην επόμενη μας συνεδρίαση, το Φεβρουάριο, να σας υποβάλω αυτές τις αδερές γραμμές του προϋπολογισμού για το 2011 και με τις δικές σας παρατηρήσεις και συνεισφορές. Ελπίζω να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Κατακλείδη, λοιπόν, ελπίζω μετά την αριστικοποίηση του εγγράφου εργασία να έχουμε ένα χρήσιμο βοήθημα που θα μας καθοδηγήσει στη δημοσιονομική διαδικασία. Ε, βέβαια θα ακολουθήσει διάλογος και με τις ε, ειδικέ επιτροπές, τις επιμέρους επιτροπές και περιμένω τα σχόλιά σας για την πρότασή μου να είναι ο κεντρικός άξονας του προϋπολογισμού το θέμα της νεολαίας, της έρευνας, κοινωνικής ένταξης και της κινητικότητας. Ελπίζω τις επόμενες εβδομάδε, να με βοηθήσετε να προετοιμάσω αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε συντόνια. Θέλει κανείς το λόγο. Monsieur, euh, Ο Σουριάν. Σας ευχαριστώ. Έχω κάποια σχόλια που θέλω να κάνω και πρώτον ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που από το Γενάρη θα αρχίσουμε ήδη να εργαζόμαστε. Αντιμετωπίζουμε νέα κατάσταση. Θα υπάρξει μία ανάγνωση για το Κοινοβούλιο. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο Μιλούμε για έγγραφο εργασία που έχει διανεμηθεί, δεν είναι ακόμη τελικό. Είμαι βέβαιος ωστόσο ότι η διαδικασία έχει προχωρήσει και νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Είναι πολύ ευνοϊκό το χρονοδιάγραμμα και επίσης είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος διότι κατά πάσα πιθανότητα ήδη τον Μάρτιο το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να διατυπώσει την άποψή του σχετικά με το τι θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον προπολογισμό. Με το νέο σύστημα, το πρώτο σχέδιο το εκπονεί η Κομισιόν. Δεν είναι όμως αδιάφορο το εάν θα λάβει υπόψη ναι ή όχι τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη τα θέματα αυτά και μαζί με τον κύριο Πέτερλε, για παράδειγμα για την νεότητα. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η έρευνα και ανάπτυξη, όπου εκεί θα αγωνιστούμε. Και ας, μη μην λησμονούμε παραδοσιακά καθήκοντα του Κοινοβουλίου, όπως την συνοχή. Θα χαρώ ιδιαίτερα αν οι πολιτικές ομάδες μπορέσουν να με υποστηρίξουν ως εισηγητή για να κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας προς την ίδια κατεύθυνση. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι τώρα σιγά σιγά να διαγράφεται το πρόγραμμα για το 2020. Αλλά δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε λόγια, ούτε πρέπει να ξαναπέσουμε σε επαναλήψεις όπως κάναμε με το λεγόμενο πρόγραμμα της Λισαβόνας. Όλοι φαίνεται να έχουμε θαυμάσιες ιδέες. Στο μεταξύ όμως από τη στρατηγική της Λισαβόνας έχουν περάσει 10 χρόνια και δεν μπορεί κανένα να ισχυριστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ισχυρότερη οικονομία και την πιο ανταγωνιστική με την ανεργία που μας πλήττει. Χρειάζεται λοιπόν να αναπτύξουμε στόχους και η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα πρέπει να είναι γεννήτρια εκείνη που θα προωθεί ιδέες, σκέψεις για να εξεύουμε τα κονδύλια του προπολογισμού που θα επιτρέψουν να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ας είμαστε λοιπόν καινοτόμοι. Βεβαίως, τα όσα έχουμε υπολείπονται των προσδοκιών μας. Εγώ θα ήμουν ευτυχέστερος των θνητών εάν μπορούσα μετά από δέκα χρόνια να πω ότι τα όσα πετύχαμε υπερέβησαν τις φιλοδοξίες μας. Πάντως θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε σωστά τα θέματα του προϋπολογισμού 2011 και πάντως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αναμένει με ενδιαφέρον να προχωρήσουν οι εργασίες για τον προϋπολογισμό αυτό και να καταβάλουμε όλοι κοινέ προσπάθειες. Uh, η Σιδωνία καλά κάνει και δεν τονίζει πολλές προτεραιότητες, αλλά λίγες μόνο. Νομίζω ότι αυτή είναι και η πεμπτουσία του προϋπολισμού να επιλέγονται ολίγες προτεραιότητες, οι οποίες βέβαια υπονοούν ότι ορισμένες μένουν στην άκρη και δεν μπορούν όλα βέβαια τα θέματα να άγονται στο ίδιο επίπεδο προτεραιότητας. Στον επόμενο γύρο της συζήτησης θα είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ρητά τους τομείς όπου θεωρούμε όπου θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να δαπανίσουμε τόσα πολλά. Γιατί μάλλον θα έχουμε ένα προπολογισμό μηδενική βάσης και όχι να προσθέτουμε σε κάθε δαπάνη ώστε να ικανοποιήσουμε όλες τις ενδεχόμενες προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Και θα έχουμε και τη δυνατότητα στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας από τη στιγμή που αναλαμβάνουμε και περισσότερες ευθύνε και έχουμε και περισσότερη μεγαλύτερη επιρροή και νομίζω ότι μπορούμε όντως να επηρεάσουμε τον τρόπο σκέψης και εντός της Κομισιόν. Και βέβαια το γεγονός ότι εμείς διορίζουμε την Κομισιόν είναι ένα υπέρ που διαθέτουμε. Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας και σας ε, υπόσχομαι την υποστήριξη της ομάδας μου ECR. Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ τη Σιδωνία για το διορισμό της ως Γενική Συγγήτριας του Προϋπολογισμού και να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτός ο προϋπολογισμός του 2011 γιατί εντάσσεται στη νέα διαδικασία που απορρέει από τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας. Και είναι βαρισίμαντο ε, για διπλό λόγο αυτό ο προπολογισμό. Θα, θα συνδυάσει τι παραδοσιακέ πολιτικέ ένωση που είναι η περιφερειακή και η γεωργική πολιτική, που μα είναι ιδιαίτερα προσφυλή, και θα πρέπει να προβλέψει χρηματοδότηση για νέες πολιτικές, ιδιαίτερα την πολιτική του διαστήματος στα πλαίσια των βιομηχανικών πολιτικών. Θα ήθελα να τονίσω κάτι που ανέφερε και η Σιδονία, την πολιτική υπέρ των νέων. Χαίρομαι που θα είναι προτεραιότητα του προπολογισμού του 2011 οι νέοι. Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας, Σιδονία, γιατί θα... ήδη έχουμε συστήσει διακοινοβουλευτική ομάδα για την νεολαία για να επισημάνουμε την ανάγκη οριζόντιας και σφαιρικής προσέγγισης, όχι μόνο υπό το πρίσμα της ε, κινητικότητας, αλλά και της ε, έρευνας, της καινοτομίας και καλό θα ήταν να ενισχύσουμε αυτή την κινητικότητα των νέων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να διευκολύνουμε και την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι που καταστήσατε το θέμα των νέων ως προτεραιότητα του προϋπολογισμού σας. Ευχαριστώ, Νταμιά. Ο κύριος Πόρτας. Άκουσα με πολύ προσοχή τις πρώτες ιδέες της συναδέλφου, αλλά έχω κάποιες αμφιβολίες. Όχι μόνο προς την εισηγήτρια, προς την Επιτροπή μας γενικά. Αρχίζουμε τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2011, ενώ δεν ξέρουμε ακόμη τίποτα για τους πραγματικούς στόχους της ενδιάμεσης αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών που θα καθορίσουν τον προϋπολογισμό του 2011. Όχι μόνο λοιπόν δεν έχουμε μια ιδέα για το πώς θα διαμορφωθεί αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση, γιατί συμπίπτουν και τα χρονοδιαγράμματά του. αλλά και πριν τον Απρίλιο ή Μάιο δεν θα έχουμε ούτε το πολιτικό έγγραφο της ε, Ισπανικής Προεδρίας που θα δώσει ένα χρονικό ορίζοντα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής μέχρι το 2020 για τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αναπόφευκτα ο προϋπολογισμός του 2011 θα είναι ένας ε, ε, προϋπολογισμός που θα συνεχίζει τους προηγούμενους. Και θα πρέπει από αυτή την ε, προϋπόθεση να ξεκινήσουμε, γιατί αν ξεκινήσουμε με διαφορετική βάση, δεν πρόκειται να τελεσφορήσουν οι προσπάθειές μας. Μέσα, στα μέσα της διαδικασίας θα διαπιστώσουμε μεγάλη διαφορά μεταξύ των αγαθών προθέσεών μας και της στιγμής πραγματικότητας. Οπότε είμαι πεπισμένος ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν είναι καθόλου καινούριος, αλλά η συνέχεια των προηγούμενων. Οπότε, πού έγινε οι αλλαγές. Ο κύριος Μπόκρος είπε ότι χρειάζονται άοκνες προσπάθειες τους επόμενους μήνες και σκληρή δουλειά τηρώντας το, τη λογική των ε, περιττών δαπανών ή των μη αναγκαίων εξόδων. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για να καθορίσουμε τους ε, λιγότερο ή περισσότερο γενναιόδωρους στόχους μας. Οπότε θα ήθελα το έργο μας για τον προϋπολογισμό του 2011 να επικεντρωθεί στις ε, δαπάνες και στο πού θα κάνουμε κάποιες οικονομίες για ανακατανομή των κονδυλίων. Τώρα, τελευταία παρατήρηση για τους νέους. Στην Ιταλία, νέοι θεωρούνται όσοι είναι μέχρι 39 ετών και ζουν ακόμη στο σπίτι των γονιών τους. Και το 80% αυτών είναι μέχρι 39 ετών. Στη Γεωργία, νέοι είναι οι νέοι Γεωργοί μέχρι τα 40 τους. Όταν μιλούμε για νέους, ποιους νέους έχουμε στο μυαλό μας. Μία πρόταση κάνω προς τη συνάδελφο. Θα πρέπει όταν χρησιμοποιούμε κάποιες έννοιες να αρχίζουμε να τις προσδιορίζουμε πρώτα. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε, για να είναι εύκολη η συζήτηση και η επικοινωνία μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Γκοντουμάνης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη συνοχή. Ο κύριος Σουριάν μας το εξήγησε. Σήμερα στην Επιτροπή Περιφερειών ακούσαμε τα σχέδια για το 2010 και την εφαρμογή το 2009 και τα οικονομικά της ε, περιφερειακής πολιτικής συνοχής. Δυστυχώς ερωτήσεις κάναμε, αλλά απαντήσεις δεν λάβαμε, σαφείς τουλάχιστον. Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειών μας ενημέρωσε ότι τα σχέδια πήγαν πολύ καλά, μάλιστα υπήρχε απορρόφηση μέχρι 99% μερικές φορές. Αλλά δεν ήταν σαφές πόσα κονδύλια μεταφέρθηκαν για το 2010 και για τον προϋπολογισμό του 2010 σε ό,τι αφορά ε, πληρωμές με βάση προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικέ του 2000-2006 γιατί αναφέρθηκαν ότι περίσσεψαν κάποια δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε είναι κάπως ε, ομιχλώδες το τοπίο, όχι μόνο από οικονομική αλλά και από πολιτική άποψη. Προσοχή λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση των πληρωμών θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ταμεία. Πολύ φοβάμαι ότι το 2011 θα βιώσουμε το τέλος κάποιων αντισυγκυριακών πολιτικών. Οπότε οι κυβερνήσεις δεν θα διαθέτουν αρκετά κονδύλια για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις. Γιατί θα πρέπει να περικόψουν τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα. Οπότε θα σκηθεί πίεση για τη χρήση, μεγαλύτερη χρήση κοινοτικών κονδύλιων, ακόμη και στην περίπτωση των διαρθρωτικών ταμείων. Η τελευταία πρόταση που καλούμαστε να συζητήσουμε είναι η πρόταση του Συμβουλίου που κάνει μία διόρθωση της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση στις περιφέρειες. Οπότε οι χώρες που θα έχουν επιβράδυση του ΑΕΠ άνω του 10% στο 2009 σε σχέση με το 2008 θα δικαιούνται περισσότερες προκαταβολές από το Ταμείο Συνοχής. Μέχρι στιγμής δεν έγινε, τέτοια, δεν έγινε έγκριση της πρότασης αυτής, θα πρέπει να την επικυρώσει το, Κοινοβούλιο. Οπότε αρμόδια κατ' ουσία επιτροπή για το θέμα αυτό θα είναι η Επιτροπή Περιφερειών που θα επιληφθεί, αλλά καλό θα ήταν να συζητηθεί και εδώ, γιατί θα έχει επιπτώσεις στο μέλλον σε ό,τι αφορά την κατανομή αυτών των κονδύλιων. Τέλος. Η κατάσταση με την κρίση είναι σοβαρή. Έχουμε και το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και πολλές νέες προτάσεις. Αλλά δεν υπάρχει πηγή για τα κονδύλια αυτά. Δεν υπάρχει ξεχωριστή δημοσιονομική γραμμή στον προπολογισμό για τα κονδύλια αυτά. Οπότε, μόνο να ελπίζουμε μπορούμε ότι θα βρεθούν κονδύλια αχρησιμοποιητά από άλλες δημοσιονομικές γραμμές για να χρηματοδοτήσουμε το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Και το ίδιο ισχύει και με άλλα ταμεία που δεν χρηματοδοτούνται άμεσα από δημοσιονομικές γραμμές του προϋπολογισμού. Και αυτό είναι σοβαρό και αντιφατικό. Πώς να αυξήσουμε τα κονδύλια αυτά απλώς με την ελπίδα ότι θα, δεν θα χρησιμοποιηθούν κονδύλια από άλλες δημοσιονομικές γραμμές, ότι δεν θα απορροφηθούν και άρα θα περισσέψουν για να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα ταμεία. Αυτό θα πρέπει να το διευθετήσουμε γιατί θα, αλλιώς στο μέλλον θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Ευχαριστώ. Merci, mon cher collègue. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Καμπάλιο. Θα ήθελα να υποστηρίξω την πρόταση στη Σιδόνια για προτεραιότητα στην παιδεία, την νεολαία, την επιστημονική έρευνα, την καινοτομία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τις επενδύσεις. Είναι πολύ σημαντικές προτεραιότητες για το μέλλον μας, για την ανταγωνιστικότητά μας. Χρειαζόμαστε νέες πηγές οικονομικής ανάπτυξης που θα στηρίζονται στην καινοτομία. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια αποδοτικότητα και των ενεργειακών, του ρηκτού πλούτου. Η αποδοτικότητά τους είναι σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης. Γι' αυτό και το θέμα της αποδοτικότητας των πόρων ε, είναι άρρηκτα δεμένο με την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού και της επιστηστικής ασφάλειας, καθώς και της αηφόρου ανάπτυξης. Και όλα αυτά τα θέματα θα είναι πολύ σημαντικά από τον προϋπολογισμό του 2011. Επίσης σχετίζονται άμεσα και με την καινοτομία και την τεχνολογική και την επιστημονική έρευνα. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Γαβριά Έχω και εγώ κάποια σχόλια για το έγγραφο εργασία ε, της συγγήτρια για την δημοσιονομική διαδικασία μετά τη θέση ισχύ τη συνθήκη της Λισαβόνας. Μόλις πριν από λίγο έλαβα το έγγραφο και μια ματιά πρόλαβα να ρίξω μόνο. Αλλά από ό,τι βλέπω, στη νέα διαδικασία που θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε μετά τη θέση ισχύ της συνθήκη Λισαβόνα. Έχουμε συγκεντρώσει σχεδόν το περισσότερο έργο το Σεπτέμβριο. Το σχέδιο προϋπολογισμού θα το έχουμε το Μάιο, γιατί δεν προβλέπεται πια προσχέδιο, κατευθείαν το σχέδιο προϋπολογισμού. Για το Μάιο όμως. Γιατί λοιπόν να μην χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε για να κάνουμε μια προεργασία, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι άλλες επιτροπές γιατί και άλλες επιτροπές θα υποβάλουν γνωμοδοτήσεις και τροπολογίες στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Έστειλα στον κύριο Σούριαν, το συνεισηγήτη, και σε εσάς πρόεδρε και σε συναδέλφους, ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια, για να έχουμε περισσότερο χρόνο και στις υπόλοιπες επιτροπές. Γιατί αυτό που ζητούμε πάντα είναι μια ευρυθή πολιτική συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Καλό θα είναι λοιπόν να κάνουμε την προεργασία έγκαιρα, ώστε το Σεπτέμβριο να έχουμε μια άνεση χρόνου. Να μην τα αφήσουμε όλα για το τέλος. Επαναλαμβάνω, δεν διάβασα ακόμη με προσοχή το έγγραφο εργασίας. Πάντως, πιστεύω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τη θέση ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα και μια και το σχέδιο προπολογισμών θα υποβληθεί το Μάιο, μπορούμε να έχουμε υπόψη αυτό το χρονοδιάγραμμα για μια καλύτερη κατανομή των εργασιών, για να μην τα αφήσουμε όλα για το τέλος, για το Σεπτέμβριο, οπότε μετά θα πρέπει να βιαστούμε και να κάνουμε άρον-άρον λίγο το έργο του προπολογισμού. Ευχαριστώ, Αΐντα. Η Αΐντα Καμπριαθάμπαλ, μα έστειλε πολύ ενδιαφέρουσε προτάσει για το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία. Και φαντάζομαι και η Συντόνια και ο Λάσλο θα συζητήσουμε την ΑΕΝΤΑ και να συνεννοηθούν ε, για κοινέ προτάσει. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τα μέλη τη Επιτροπή, ε, γιατί το έγγραφο εργασία τη Συντόνια μόλι σήμερα καταφέραμε να το μοιράσουμε. Οπότε όλοι το λάβαμε με την έναρξη της συνεδρίασης. Στο παράρτημα υπάρχει ένα σχέδιο χρονοδιαγράμματος μέχρι τον Νοέμβριο του 2010 για την έγκριση του προπολογισμού του 2011 και έχετε και ένα σύντομο πίνακα που μοιάζει με κινούμενο σχέδιο. Μόνο ε, πρόσωπα λοιπόν που εξηγεί τη νέα διαδικασία που μας εξήγησαν η Συντόνια και άλλοι. Έχουμε μία ανάγνωση πια, οπότε κάθε κοινοτικό θεσμικό όργανο θα πρέπει να θετήσει θέσεις τακτικής και με μεγαλύτερη σοβαρότητα να καταλήξει και να ανακηρύξει τις πολιτικές του επιλογές. Επίσης, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χρόνο που θα έχουμε στους πρώτους μήνες του χρόνου για να προπαρασκευάσουμε την πολιτική μας θέση σε συνεργασία με τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Και ο Γκέρον Φέρμαν, ο τελευταίος ομιλητής. Thank ε, Κάποια σχόλια. Καταρχήν να συγχαρώ τη Μαθηδόνια που ορίστηκε εισηγήτρια. Ήμουν εισηγητής για τον προπολογισμό πριν από 8 χρόνια και είναι πολύ ωραία εμπειρία. Ελπίζω να, ε, είναι το ίδιο, να ισχύσει το ίδιο και για σας. Τώρα όσον αφορά τον ε, σχεδιασμό και αυτό το έγγραφο εργασίας, δεν πρόλαβα να το ρίξω μια μάτια αλλά να σχολιάσω περισσότερο κάτι που απευθύνεται στον πρόεδρο της Επιτροπής και όχι στην εισηγήτρια, γιατί εκτός των όσων έχουμε εδώ σε αυτό το πίνακα έχουμε πολλά περισσότερα. Δηλαδή, έχουμε ολόκληρη την υπόθεση της διαθεσμικής συμφωνίας του δημοσιονομικού κανονισμού, χρηματοπιστωτικού κανονισμού, έχουμε ένα σώρο άλλε συζητήσει που επεμπίπτουν στι εντολέ τη Επιτροπή μα και γενικά θα θέλουμε έναν συνολικό προπολογισμό για όλο το χρόνο για την Επιτροπή μα. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί θα είναι ένα πολύ δύσκολο έτο για την Επιτροπή μα. Ο προπολογισμό του 2011 είναι βεβαίω το κεντρικό τμήμα, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει ταυτόχρονα να κάνουμε. Ο πρόεδρο λοιπόν και η Γραμματεία θα πρέπει να μα δώσουν όχι μόνο το σχεδιασμό για τον προπολογισμό, αλλά και γενικότερα για τη δουλειά όλου του χρόνου, να το προγραμματίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά τη συζήτηση για τι κατευθυντήριες γραμμέ, Εγώ συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν. Δηλαδή, θα πρέπει να, πάρουμε, να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία και να προσπαθήσουμε εμεί να ορίσουμε την ημερήσια διάταξη. Αλλά επίση είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσπαθήσουμε να ε, φτιάξουμε ένα συμπυκνωμένο ε, γραφό, όχι ένα μεγάλο μακροσκελές κείμενο με 79 παραγράφους, γιατί θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να κερδίσουμε την μάχη με το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να έχουμε μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου μαζί με την πλευρά μας. Και αυτό σημαίνει ε, προηγούμενη βάθος συζήτηση μεταξύ μας. Και να αναφέρω και το εξή που επίσης θα πρέπει να κάνουμε, δηλαδή μια ανάλυση των προβλημάτων που είχαμε φέτος. πάση περιπτώσει τον περσμένο χρόνο για το 2010, για τον προπολογισμό του 2010, γιατί αυτά μας ακολουθούν και για τον επόμενο χρόνο. Και θα χρειαστεί και τουλάχιστον δύο από αυτά τα έχουμε στην ατζέντα για σήμερα. Δηλαδή τα ανώτατα όρια για την κατηγορία 1α που έχουμε πολλέ από τι προτεραιότητε μα για την κοινωνική ένταξη, την πολιτική για το διάστημα κτλ. Και δεν υπάρχει χώρο για όλα αυτά. Θα πρέπει πραγματικά πολύ νωρί να κάνουμε μια στρατηγική σημασία συζήτηση για το πώ θα χειριστούμε αυτό το πρόβλημα. Και όπω είπα, θα γίνει αργότερα σήμερα στην έκθεση του κυρίου Άμπαντ για το GMES. Αλλά έχουμε και την κατηγορία 5 που έχουμε και επίση στην ημερησία διάταξη και συνδέεται όχι μόνο με, αριθμητικά, με τα στοιχεία τα αριθμητικά, αλλά και τι διοργανικέ σχέσει την Συμφωνία Κυρίων, το όριο 20% για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στην κατηγορία 5 που σήμερα είναι μια τελείως και νέα κατάσταση και θα πρέπει να το συζητήσουμε νωρίς, γέρος, ώστε να μην ε, αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για τις ε, διοργανικές σχέσεις. Γιατί όλα αυτά δεν αφορούν την συνηθισμένη συζήτηση για την κατηγορία 5. Έχουμε τώρα συζήτηση για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Έχουμε συζήτηση για τους μεταβατικούς κανόνες, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον προπολογισμό του 2011, τις μεταφορές κτλ. Και έχουμε και ένα σωρό συζητήσει που σχετίζονται με την διοργανική συμφωνία και τις ε, σχέσεις. Μερικά πράγματα που πρέπει να τα λύσουμε λοιπόν όσο γίνεται πιο σύντομα, να υπάρξει μια στρατηγική συνεννόηση ανάμεσα στι ομάδε για να αντιμετωπίσουμε τον προπολογισμό του 2011. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Εγώ θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να χαιρετήσω την Κατρίν Κικιά που ήταν η προκάτοχό σα και που είναι παρούσα στην αίθουσα. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση. Αν ήρθε να δει πώς ε, και αν μένουμε πιστοί ή άπιστοι στην πολιτική της κληρονομιά, πάντως έχει μια άποψη πολύ παράξενη για την ε, πίστη, γιατί κάθεται στην ομάδα των, στις θέσεις της ομάδας των εμπειρογνωμόνων της EFD. Καλώς ήρθες ε, αγαπητή Κατρίνα. Τώρα, ε, ο Γκέρχαν ε, τόνισε πολύ σημαντικά σημεία. Όντω θα πρέπει όσο γίνεται πιο σύντομα να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα συνολικό, πλήρε. Όχι μόνο πράγμα που ήδη ισχύει για την ετήσια διαδικασία του προπολογισμού, αλλά και για τα άλλα κείμενα ή αποφάσεις που είναι σημαντικά και που μας περιμένουν. Εργαζόμαστε επί αυτού. Είναι κάπως δύσκολο να είμαστε συγκεκριμένοι από τη στιγμή που δεν έχουμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να έχει αναλάβει. Ξέρουμε ποιος θα είναι υπεύθυνο για τον προπολογισμό, αλλά ο ίδιος δεν έχει ακόμα αναλάβει καθήκοντα και για μερικά από τα πιο σπουδαία κείμενα η επιλογή του χρονοδιαγράμματος όσον αφορά την ευθύνη της Κομισιόν δεν εξαρτάται από εκείνον μόνο, αλλά είναι σαφές ότι θα μεριμνήσουμε ώστε να έχουμε αυτές τις διευκρινήσεις, να μπορέσουμε να δουλέψουμε όσο γίνεται από καλύτερε συνθήκες. Ο Γκέρχαν επίσης σωστά θύμισε ότι για το Κοινοβούλιο Οι νέε ευθύνε που μα δίνει η συνθήκη τη Λισαβόνα καθιστούν ακόμα πιο απαραίτητοι την ε, όσο δυνατόν ευρύτερη πλειοψηφία. Θα θυμάστε πως το καταφέραμε σε αυτό το πνεύμα να υιοθετήσουμε τον προπολογισμό 2010 με πλειοψηφία των 4 πέμπτων των εκπεφρασμένων ψήφων. Άρα λοιπόν πολύ πάνω από τα δυο τρίτα. Ήταν ένας πολιτικός στόχος που είχαμε ορίσει για να σηματοδοτήσουμε την ισχύ μας απέναντι στα άλλα θεσμικά όργανα. Και νομίζω πως με αυτό το πνεύμα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Και έτσι μάλιστα το παρουσίασε και η Σιδονία. Και γι' αυτό και θελήσαμε από σήμερα να γίνει και όλα σε αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τις ε, πρωτοβουλίες και τις ανησυχίες των όλων μας. Μια επιφανειακή πρώτη ανταλλαγή απόψεων ένας πρώτος γύρος, αλλά είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε από την αρχή του χρόνου να, με τις, την καλή συνήθεια να συνεργαζόμαστε. Η Επιτροπή μας το κατάφερε να το κάνει και τα προηγούμενα χρόνια και θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα τα επόμενα χρόνια. Επίσης, ακούγοντας σας ε, για, νο, ίσως ο Χάιμερ ε, μέσα στο πλαίσιο των ευθυνών του ως μόνιμος ε, εισηγητή για τι δημοσιονομικέ προοπτικέ να μπορούσε να μα κάνει ένα σύντομο έγγραφο εργασία, έναν πίνακα για το απερθώρια που υπάρχουν ακόμα ανακατηγορία και αναυποκατηγορία. Για την αλήθεια ότι μετά από τις διαπραγματεύσεις που είχαμε για τον προϋπολογισμό 2010 τα περιθώρια ε, περισσότερο σε λεπτά τα μετράμε παρά σε εκατομμύρια ευρώ. 0,01 ίσως να υπάρχει και κάποιο μικρό περιθώριο ακόμα. Λοιπόν, κύριε Συγχύτρια. Α, ναι, Χάιμερ. Α, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Ο Χάιμερ για αυτό το σημείο και μετά ο κύριος Κολίνο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να συνεχίσω από αυτά που ανέφερε πριν ο κύριος Φραμ βρίσκονται μπροστά μας μήνες με πολλή δουλειά. Τώρα, εάν θα είναι δύσκολο αυτό το έτος από άψη προϋπολογισμού, θα εξαρτηθεί από τον ζήλο με τον οποίο η Κομισιόν θα κάνει προτάσεις σεβόμενη τη διαθεσμική συμφωνία. Και κατά πόσον θα ληφθούν υπόψη τα πράγματα που έχουμε ήδη πει σε διάφορα ψηφίσματα, ξεκινώντας από την συνθήκη τη Λισαβόνα με την έκθεση τη Καθήν και τα όσα είχαμε πει για την αναθεώρηση του προπορισμού υπό δική μου τότε ε, διεύθυνση και τα όσα είπαμε και με τον Λάσλο Σούριαν τον Δεκέμβριο. Θα εξαρτηθεί βέβαια σε μέγα βαθμό και γι' αυτό ο Δεκέμβριο υπήρξε τόσο σημαντικός για το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες, εξετάσουμε δηλαδή ότι και τον προϋπολογισμό 2011 η πολιετή συμφωνία που θα χρειαστεί να θεσπίσουμε θα έχει σημαντική επιρροή και σε σημαντικές κατηγορίες και γραμμές του προϋπολογισμού. Το ερώτημα που μένει είναι τι περιθώριο μας μένει και η απάντηση είναι εύκολη σχεδόν καθόλου. Ή εάν θέλετε θα πρέπει να ψάξουμε απελπισμένα ή αδίποτε περιθώρια ή να κάνουμε μεταφορές από κατηγορία σε κατηγορία. Πράγματα που κάναμε στο παρελθόν με αρκετή επιτυχία, αλλά πάντως τα διαθέσιμα περιθώρια δεν είναι αυτά τα οποία είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτά τελειώνουν. Και γι' αυτό και το ενδιαφέρον ερώτημα και σε σχέση με τα όσα θα συζητήσουμε με τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές για τον προπορισμό 2011 και εγώ θα υποβάλω σχετικό έγγραφο στις επόμενες συνεδριάσεις τι θα κάνουμε με την προσαρμογή της διαθεσμικής συμφωνίας διότι προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της διαθεσμικής συμφωνίας και αυτό γίνεται αποκλειστικά μεταξύ των θεσμικών οργάνων θα ήθελα να ανακοινώσω ήδη στους συναδέλφους ότι εάν δεν μας αρέσουν τα όσα θα ακούσουμε, θα πούμε όχι. Θα χρειαστεί να συζητήσουμε και πώς θα κατανείμουμε αυτή την τροποποίηση. Εάν πούμε ότι ένα μέρος της διαθεσμικής συμφωνίας θα περάσει στο, στην νομοθεσία με γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, είναι τεχνικής ε, φύσεως προσαρμογή αυτή ή προκύπτει από την προσαρμογή των πολιτικών προτεραιοτήτων λόγω Λισαβόνας. Και μήπως προκύπτει και ως ανάγκη ενός δημοσιονομικού δελτίου από την ε, πυραμίδα του οργανογράμματος μέχρι την εξωτερική υπηρεσία, μέχρι θέματα ε, διαστημικής συνεργασίας κλπ. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε όταν Φεβρουάριο-Μάρτιο θα υποβάλει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν γίνει τέτοιοι υπολογισμοί. Υπάρχει ένα facing in, μια σταδιακή εισαγωγή. Έχουμε να περιμένουμε ορισμένα πράγματα. Ή προωθούνται όλα προς την κατεύθυνση του 2020. Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Καθώς επίσης και το ερώτημα, τι θέλουμε ως Κοινοβούλιο και εκκινώντας από την υφιστάμενη διαθεσμική συμφωνία, να περάσει στην, στον δημοσιονομικό κανονισμό, σε διαδικασία συναποφάσεως δηλαδή, και τι θέλουμε να παραμείνει μέσα στην υποπολιτική διαπραγμάτευση διαθεσμική συμφωνία. Ορισμένα πράγματα καταργούνται, είτε υποχρεωτικά είτε μη υποχρεωτικά. Υπάρχουν κεφάλαια που κατά τη γνώμη μου πρέπει να ανοίξουν απολύτως. Θυμούμε πώς διαπραγματευτήκαμε το δικαίωμα ενημέρωση του Κοινοβουλίου για την ΚΕΠΑ. Το κατακτήσαμε το δικαίωμα αυτά, αυτό. Η διαβούλευση αυτή, κρίνω εγώ, τη λειτουργεί αρκετά καλά. Αλλά δώσαμε και εμείς κάτι. Δηλαδή να μην δημιουργούμε για παράδειγμα αποθεματικά σε αυτές τις γραμμές του προπολογισμού και ορισμένα άλλα. Τώρα όμως είναι και η σειρά των συνομιλητών Και επομένως όλο το κεφάλαιο για την ΚΕΠΑ και την πολιτική Άμυνα πρέπει να είναι εκ νέου αντικείμενο διαπραγμάτευση και να προσαρμοστεί. Εξού προκύπτει κιόλα ότι αυτό πρέπει να γίνει παραλίλω με την σύνταξη της νομοδότησης για τη δημιουργία της εξωτερικής υπηρεσίας η οποία θα προέλθει ως επί έκθεση από την Συνταγματική Επιτροπή για να μιλούμε με μία φωνή και για να κάνουμε και την απαραίτητη προσαρμογή της διαθεσμικής συμφωνίας, ώστε και με αυτήν και με τον δημοσιονομικό κανονισμό να μπορούμε να συνεπηρεάσουμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Θα εξαρτηθεί κατά μέγα βαθμό η κίνηση αυτή από το τι θα υποβληθεί από πλευρά τη Κομισιόν. Εάν θα θεωρήσει η Κομισιόν ότι βρίσκεται σε θέση εν ώψη και τη μελλοντική εξελίξεως της ε, χρηματοδοτήσεω να δώσει κάποιες πρώτε κατευθύνσει. ή αν θα χρειαστούμε να το κάνουμε εμείς. Και σε παλαιότερες διαπραγματεύσει. υπήρξαν υπήρξαν περιπτώσεις όπου, όπου, όπου οι συνομιλητές μας δεν τολμούσαν να καταθέσουν νούμερα και τότε κινηθήκαμε πρώτοι εμείς. Αυτά ήθελα να πω και προς την εισηγήτρια απαντώντας λίγο και σε αυτά που είπε ο Γκόραν Φάρμ και όταν ενδεχομένως θα κάνει στις 17 του επόμενου μηνός η Κομισιόν βέβαια είναι και δύσκολο αυτό για την νέα Κομισιόν γιατί η προεργασία έχει γίνει ήδη υπό ευθύνη της απερχόμενης Κομισιόν και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα δράσει η νέα Κομισιόν εφόσον περιοριστεί μόνο στο τεχνικό και δεν κάνει πολιτικές προσαρμογές, πώς θα συνεννοηθούμε με τον νέο Επίτροπο και με τους άλλους συναρμόδιους Επιτρόπους και θα κάνουμε τις απαραίτητες πολιτικά συζητήσεις ώστε να πετύχουμε το δυνατόν πιο έγκαιρα την σύναψη αυτής της διαθεσμικής συμφωνίας. Αλλά αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος διότι και μέχρι το φθινόπωρο η Κομισιόν μπορεί να κάνει προτάσεις προσαρμογής για τη διαδικασία του προπολογισμού και νούμερα τα οποία θα χρειαστεί να συζητήσουμε ακόμη μέσα στο 2011. Άρα ο χρόνος είναι ουσιώδης παράγοντας, αλλά αυτό που μετρά είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα για το 2011. Θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε να καταθέσω ορισμένες σκέψεις για την επόμενη συνεδρίαση ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια πράγματι εντατική συζήτηση. Ευχαριστώ, Ράιμερ. Πολύ εύστοχα τα σχόλιά σου. Ο κύριο Κολίνο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ πω δεν είναι θέμα χρονοδιαγράμματος, αλλά θέμα στόχων που πρέπει να επιτευχθούν. Ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο Σιδόνια για το πώς ε, ιεράρχησε τις πρωτοβουλίες για το 2011. Θα, το πρόβλημα της νεολαίας ε, των φοιτητών, των ερευνητών, ε, κοινωνική ένταξη, σημαίνει αυτό πως θέλουμε σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή, θέλουμε να ερμηνεύσουμε και πλέον έχουμε και τον ε, προϋπολογισμό με βάση τη Λισαβόνα, θέλει να ερμηνεύσει την κοινωνική εξέλιξη στην Ευρώπη. Προηγουμένως ο συνάδελφος Πόρτα στην παρέμβασή του θύμισε πως στην Ιταλία είναι κανείς νέος μέχρι τα 39. Εγώ ω Ιταλό δεν συμφωνούσα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή στην Ιταλία γίνεται τώρα μια κοινωνική συζήτηση, κοινωνιολογική συζήτηση για την εξέλιξη τη κοινωνία και τη οικογένεια και για την εξέλιξη του προβλήματο όταν οι νέοι φεύγουν από το σπίτι. Τη στιγμή δηλαδή που οι νέοι φεύγουν από το σπίτι του, πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι ο κοινωνικό αντίκτυπο όσον αφορά το πρόβλημα τη κατοικία, το ε, ε, πρόβλημα του νέου οικογενειακού πυρήνα και ούτω κάθεξή. Το να ασχοληθούμε λοιπόν με το θέμα της νεολαίας μέσα στον προπολογισμό του 2011 ε, και από όλε αυτές τις απόψεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι ακόμα, ένα σημείο το οποίο παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή και αφορά τους νέους σε θέματα της ε, Επιτροπής Μεταφορών, αφορά την ασφάλεια, την οδική, την οδική συμπεριφορά που συνδέεται με τις συνήθειες ιδιαίτερα των νέων, γιατί γνωρίζουμε ότι από τις συμπεριφορές ε, γεννιέται μια καλή κοινωνία και οι νέοι είναι η κληρονομιά της Ευρώπης, ε, άρα λοιπόν είναι μια πτυχή την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο. Είναι ένα πολιτιστικό θέμα, θέμα αξιών, θέμα συμπεριφορών. Πολύ συχνά οι νέες γενναίες ε, όσο, που είναι πιο κοντά σε ληστικές πτυχές της ζωής και ξεχνούν αυτού του είδους της ε, συμπεριφορές. Το γεγονός επίσης ότι εμείς ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο προβλέπουμε κάποιες χαρακτηρίες γραμμές για τον προπολογισμό 2011 θα πρέπει να το δούμε με θετικό τρόπο. Δεν είναι αρνητικό γιατί τον μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι θετικό. Ε, επίσης τώρα όσον αφορά τους στόχους 2020 και τις δαπάνες για τις οποίες μιλήσαμε και πριν, εγώ πιστεύω πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι εξαιρετικά σταθερό στις απόψεις του. Εμείς είμαστε εκπρόσωποι των λαών και σίγουρα όχι η γραφειοκρατία. Ούτε η εθνική ούτε η ευρωπαϊκή. Από εμά εξαρτώνται οι πολιτικέ γραμμέ, από εμά εξαρτώνται οι κατευθύνσει προ τι οποίε οι πολίτε έπειτα θα... από τι οποίε έπειτα οι πολίτε θα κάνουν τι επιλογέ του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Σε ό,τι αφορά την ηλικία, στην ε, Γαλλία ήμουν κάποτε σε ένα κόμμα που όπως όλα τα πολιτικά κόμματα έχει και μια πτέρυγα νεολαία. Και για να ενταχθεί κανείς ε, στο τμήμα τη νεολαία ή θα έπρεπε να είναι κάτω των 30 ετών, είτε να ήταν κάποτε κάτω των 30 ετών. Οπότε, ε, στην επαγγελματική σταδιοδρομία, στην πολιτική σταδιοδρομία για ένα μεγάλο διάστημα μας έλεγαν είστε πολύ νέος και κάποια στιγμή μας είπαν δεν είστε αρκετά νέος, είστε πολύ ηλικιωμένο πια. Λοιπόν, Σιδόνια, ποια είναι η γνώμη σου μετά αυτή την πλούσια συζήτηση. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω θερμά για όλες τις παρατηρήσεις, τη σημείωσα προσεκτικά. Η πρώτη μου εντύπωση είναι ότι υπάρχει υποστήριξη για τις αδρές γραμμές που σας παρουσίασα, κάτι που μου δίνει κίνητρα και ενθουσιασμό να συνεχίσω. Άκουσα και πολύ πιο συγκεκριμένα σχόλια. Μπορώ να αναλύσω κάποιες παρατηρήσεις. Υπάρχει χρόνος. Ναι, καταρχήν ο προπολογισμό του 2011 δεν είναι απομονωμένος. Θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα προβλήματα από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και κυρίως ε, τα σύντομα περιθώρια. Κύριε Μποκρός, δεν φοβάμαι τις περικοπές. Ιδιαίτερα όταν είναι πολύ στενά τα περιθώρια, θα πρέπει να έχουμε το κουράγιο να μπούμε σε μια διαδικασία αναθεώρησης για να δούμε πού υπήρξε ε, υποχρησιμοποίηση, υποαπορρόφηση, που έμειναν αχρησιμοποίητα κονδύλια. Όχι μόνο αναθεώρηση λοιπόν του πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά να δούμε που έμειναν ανεκμετάλλευτα κονδύλια για να τα διοχετεύσουμε αλλού. Οπότε και το θέμα της, των πηγών χρηματοδότησης με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ο κύριος Γκοντμάνης είπε ότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε ότι ορισμένε γραμμές είναι σαν πηγάδια αντλούμε από εκεί κονδύλια χωρίς να προβληματιζόμαστε γιατί είναι τόσο δαψιλώς εφοδιασμένες αυτές οι γραμμές. Και αυτό έχει σχέση με την αναθεώρηση της ε, εφαρμογής. Αλλά έχουμε και μια μονάδα παρακολούθησης. Εκεί νομίζω θα μπορούσαμε να εξετάσουμε από πού θα μπορούσαμε να βρούμε τα κονδύλια που μας λείπουν. Νέα διαδικασία. Α, και το χρονοδιάγραμμα που είναι πολύ σημαντικό. θα χρειαστεί στο χρονοδιάγραμμα να προσθέσουμε και κάποιες παράλληλες διαδικασίες. Και συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώραν Φέρμ. Αλλά θα ήθελα να έχουμε εκπρόσωπο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί θα ζητήσω και τη δική της βοήθεια και συμβολή στο χρονοδιάγραμμα. Για παράδειγμα, τι γίνεται με το έργο, με, το, με την επιστολή εκτελεστότητας. Θα, έχει, θα προλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τις τροπολογίες μας και να καταρτήσει την εκτελεστική επιστολή. Οπότε το χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί και από την συμμετοχή και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς θα εφαρμόσουμε τη νέα διαδικασία. Η Ισπανίδα συνάδελφος ρώτησε γιατί τα αφήνουμε όλα για το δεύτερο εξάμεινο. Απότερο στόχος μας είναι φυσικά να γίνει ένας ισότιμος καταμερισμός του έργου μας στον χρόνο. Και εκεί θα χρειαστώ τη συνεργασία όλων των πολιτικών ομάδων, ώστε ένα τμήμα της συζήτησης να διεξαχθεί στο πρώτο εξάμεινο. Εγώ είμαι πρόθυμη ήδη από τώρα να συνεργαστώ μαζί σας. και αν ήδη καταθέσουμε τροπολογίες από τις αρχές ε, Σεπτεμβρίου, θα περάσουμε όλο μας το καλοκαίρι με τις τροπολογίες. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος μας για τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα καθόμαστε και να συντάσσουμε τροπολογίες ε, στο κατακαλό καιρό. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε τον Αύγουστο από τροπολογίες. Πάντως θα έχω στενή συνεργασία και με τις ε, επιμέρους επιτροπές πριν τον Ιούλιο και στη διαδικασία της κατάρτισης τροπολογιών θα πρέπει να είμαστε επιθαρχημένοι και ρεαλιστικοί. Γιατί δεν προβλέπονται πια δύο αναγνώσεις, παρά μόνο μία. Οπότε μία ευκαιρία θα έχουμε. Πειθαρχία λοιπόν και ρεαλισμό τη τροπολογία γιατί δεύτερη ευκαιρία δεν θα υπάρξει. Μία και μόνο ανάγνωση και μετά κατευθείαν συνδιαλλαγή. Επίσης θα ήθελα να επιδείξουν εγκράτη και αυτοπιθαρχία και οι επιμέρους επιτροπές. Να περιοριστούν λοιπόν στις προσδοκίες τους με τις τροπολογίες. Αλλά και η Επιτροπή προϋπολογισμών θα πρέπει να δείξει μια αυτοπιθαρχία. Και προσβλέπω σε στενή συνεργασία και στη συμβολή σας. Δεν ήθελα τώρα εδώ να κάνω μια θεωρητική συζήτηση ακαδημαϊκή πότε κάποιος θεωρεί ηλικία και πότε χάνει αυτή την ιδιότητα. Το θέμα δεν είναι ποια φιλοσοφία έχει ο καθένα για τους νέους. Το θέμα είναι ότι οι νέοι είναι ένας πόρος. Είναι μια πηγή πλούτου που δυστυχώς εξαντλείται, αρχίζει και εξαντλείται αυτός ο πλούτος, αυτός ο πόρος της ευρωπαϊκή Ένωσης. Οι νέοι είναι η ευκαιρία μας και είναι ο πόρος που θα δημιουργήσει πλούτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Το θέμα δεν είναι πότε θεωρείται κάποιο νέο, αν είναι 19, 27 ή 39. Το θέμα είναι ότι ο, νέος νέο είναι ευάλωτο. Ιδιαίτερη μετάβασή του από τι σπουδέ στην εργασία είναι πολλέ φορέ ε, προβληματική. Και αυτό είναι η λέξη κλειδί. Είναι το σημείο καμπής η μετάβαση από τους ακαδημαϊκούς κύκλους, από τις σπουδές, στον επαγγελματικό βίο. Και καλό θα είναι να εξασφαλίσουμε όσο δυνατό καλύτερη παιδεία γίνεται, αλλά να ε, προσέξουμε και το θέμα της μετάβασης και της ένταξης. Γι' αυτό ανέφερα και το θέμα της κινητικότητας και τα προγράμματα που ήδη λειτουργούν όπως το Έρασμος. Και επίσης να κατανοήσουμε και να περιλάβουμε και την έρευνα, τους πανεπιστημιακούς κύκλους, την κινητικότητα των μαθητευομένων ή την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ή των επαγγελμάτων στα πλαίσια της κινητικότητας των νέων. Εγώ σπούδασα κοινωνιολογία και εργάστηκα ως κοινωνιολόγος. Αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον κλασικό αυτό κύκλο ε, σχολείο, εργασία, ε, σύνταξη. Αυτός ο κύκλος πια αλλάζει. Γιατί δεν είναι ότι κάποιο μετά τις σπουδές ε, ε, αρχίζει και δουλεύει και δεν ξαναπιάνει τις σπουδές. Τώρα ο, ο κόσμος ε, ενημερώνεται και σπουδάζει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωή. άρα κρατάει τον ενικό του χαρακτήρα, μια και ε, διδάσκεται συνεχώς. Αρχίζει και γίνεται κάτι, ένα κυκλικό φαινόμενο η μόρφωση. Και πολλές φορές είναι καλό να εξασφαλίσουμε μια κινητικότητα μεταξύ εργασία και σπουδών, γιατί μερικοί έχουν δυσκολίε να ξαναπιάσουν τι σπουδέ του ενώ εργάζονται. Κινητικότητα λοιπόν είναι λέξη κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σας ανέφερα και σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Ευχαριστούμε Συντόνια. Νομίζω ότι όλοι εκτίμησαν και τα προσόντα σας και τις ικανότητές σας και το πνεύμα που διέπει αυτή την προσπάθειά σας ε, κατάρτιση των προπολογισμών σε αυτή την κρίσιμη χρονιά. Παίρνουμε τώρα στα λοιπά τμήματα, πολύ σημαντικό στοιχείο του προπολογισμού και η Χέλγα Τρίπελ θα μας κάνει την ενημέρωση για τις πολιτικές επιλογές του 2011 στα λοιπά τμήματα. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω βέβαια γερμανικά. Θα ήθελα πρώτα με όλο τον σεβασμό που έχω στον κύριο Μπόκροφ και στις πολιτικές του επιθύσεις αν ήταν πράγματι έτσι όπως λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή πέρασε τα σημαντικά θέματα που το ενδιαφέραν και τις φιλοδοξίες του, τότε ο προπολογισμό θα ήταν πολύ διαφορετικός από αυτόν που έχουμε τώρα. Για να... Είναι σημαντικό να το πω αυτό για να δούμε τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Δεύτερη προκατακτική παρατήρηση και συμφωνώ με τον κύριο Μπέγκε, όπω μίλησε προηγουμένω. Εν ώψη και τη συζητήσεω που θα γίνει σχετικά με το ύψο του προπολογισμού του Κοινοβουλίου, συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, είναι σημαντικό να επανεξετάσουμε τη στρατηγική μα κατάσταση. Δηλαδή, τι προσφέρει η συνθήκη τη Λισαβόνας και για την Κομισιόν, αλλά και για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Τι σημαίνει δηλαδή για αυτά και κατά πόσο θα είμαστε επιτυχείς βέβαια στην εφαρμογή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ωστόσο, χρειαζόμαστε πρώτα μια πολιτική συνεννόηση σχετικά με το ότι ναι μεν πετύχαμε τώρα να τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας, ωστόσο έχουμε κοινό συμφέρον να την εφαρμόσουμε και να προσαρμόσουμε τους τρόπους εργασίας μας στο περιεχόμενό της. Και σε ό,τι αφορά το έργο μας ως κοινοβουλευτικών ανδρών και γυναικών, αλλά και την εργασία των επιτροπών και τον τρόπο εργασίας άλλων υπηρεσιών από, τα πολιτικά, από τις ε, πολιτικές υπηρεσίες μέχρι τη βιβλιοθήκη. Εάν εξετάσουμε τον εξοπλισμό που διαθέτει το Αμερικανικό Κογκρέσο και εμείς, δεν μπορεί να κάνει κανείς σύγκριση ένα προς ένα, αλλά ο εξοπλισμός μας, ευρία ενία, είναι ακόμα πάρα πολύ μετριόφρονο θα το πω έτσι, απέναντι στον Αμερικανικό. Μέχρι τώρα έχουμε συμφωνήσει ότι ο προπολογισμό του Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20% και πάντως όχι στο έτος 2010. Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για Parliament's Agreement που όταν γεννήθηκε αυτή η απόφαση αυτά τα 20% ήταν χωρίς η διεύρυνση, χωρίς πολιτική κινήτων και χωρίς καθεστώς των ευρωβουλευτών. Πέρσι όμως πάλι 20% αλλά συμπεριλαμβάνουν όλων αυτών των παραγόντων που μόλις ανέφερα. Ε, μπορεί κανείς να πει λοιπόν ότι υπερβήκαμε τα όσα διαθέταμε. Πρέπει λοιπόν να εγκύψουμε σε μια στρατηγική συζήτηση για το τι σημαίνει η Λισαβόνα και τι μπορούμε να αναμένουμε από αυτήν. Δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι ξοδεύουμε παραπάνω από όσα διαθέτουμε, α το πω έτσι. Συζήτησα με τους συνεργάτες μου τι θα σημαίνει αυτό για το προπολογισμό του 2011, προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Θα πω τώρα στα αγγλικά αρχίζοντας με το 30% παραδοσιακό για, την, για τον τίτλο 5. και το τι θα σημάνει, για παράδειγμα, η πολιτική ακινήτων κλπ. Βασιζόμενοι σε μια προβολή των προβλέψεων για το 2010 ε, και 2011, θα οδηγηθούμε σε έξτρα δαπάνες ύψους 22,2 εκατομμυρίων ευρώ. Εάν διατεθεί, εάν ε, ε, ε, παραμείνει το ποσό για τον κάθε ευρωβουλευτή, συν τα 3.000 ευρώ, τα οποία συζητούνται ακόμα, που σημαίνει ότι θα χρειαστούμε ακόμα 35,49 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ όμω συνδέεται και ένα άλλο θέμα. Εάν διαθέτουμε περισσότερο προσωπικό ή αν μας διαθέσουν περισσότερα χρήματα για περισσότερο προσωπικό, πρέπει βέβαια να δεχθούμε ότι η συνέπεια θα είναι τι γίνεται με τα υπόλοιπα, δηλαδή τι κάνουμε με τα ακίνητα. Πρέπει να τροποποιήσουμε όλη τη διάθρωση των, ακινήτων μας αυτά είναι εκτό νέων ακινήτων. Τι σημαίνουν αυτά για την εργασία μα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά είναι σαφέ ότι αυτά τα πράγματα συνδέονται. Δεν είναι μονάχα η ανάγκη να εντοπίσουμε νέα χρήματα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα καθημερινά προβλήματα τη δουλειά μα. Η δεύτερη ερώτηση που προκύπτει τώρα για την αύξηση των αμοιβών και τι θα σημαίνει. Τα καθυστερούμενα εκτιμούνται σε 1,085% και για ένα αριθμό μηνών του 2010 θα είναι 245 εκατομμύρια για όλες τις, για θεσμικά όργανα και 14 εκατομμύρια μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, τα δύο αυτά ποσά μαζί και σύμφωνα με την συνηθισμένη αύξηση από 2010 σε 2011 του τίτλου 5 φτάνουμε στα 51,2 εκατομμύρια. Και αυτά τα δύο ποσά, εφόσον προστεθούν σημαίνουν ότι χρειαζόμαστε λίγο πολύ αυτό το ποσό για την εφαρμογή αυτής της νέας στρατηγικής. Άρα δεν έχουμε περιθώριο, δεν μας παραμένει περιθώριο. Και το άλλο πράγμα που πρέπει να συζητήσουμε ή τέλο πάντων να εκτιμήσουμε, να λάβουμε υπόψη, είναι ότι υπάρχουν νέες πληροφορίες ότι ίσως θα υπάρξει επιστροφή 85 εκατομμυρίων από την βελική κυβέρνηση, χρήματα δηλαδή τα οποία ξοδέψαμε από τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου για τη διαμόρφωση του, ε, περιφερειακού, του περιμετρικού χώρου γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ίσως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια αξίωση επιστροφής και μπορούμε να βασιστούμε σε αυτήν εφόσον βέβαια μας επιστραφούν αυτά τα έξτρα χρήματα. Κάτι το οποίο θα επηρεάσει βέβαια το 20% και αν θέλουμε να το διατηρήσουμε και αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το 20% τότε θα υπάρχει κάποιο περιθώριο. Από την άλλη μεριά, και αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα που θέτω, είναι το στρατηγικό ερώτημα δηλαδή, εάν παραμένουμε σε αυτά τα 20% και για πολιτικούς βέβαια λόγους, σημαντικούς πολιτικούς λόγους, η εργασία μας και για να μπορέσουμε να εργαστούμε καλά και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που θέτει η συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχουν ορισμένα επιχειρήματα που λένε ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Και ένα ακόμα θέμα, η ομάδα μου των Πρασίνων θα ήθελε ως μέρος του προϋπολισμού του Κοινοβουλίου εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε λίγο πολύ παντού Microsoft. Όμως αναπτύσσεται η ψηφιακή αγορά και ε, αγωνιζόμαστε κατά αυτού του μονοπωλίου μιας μεγάλης εταιρείας η οποία προσφέρει μόνο πρόσβαση στα δικά της ε, λογισμικά και θέλουμε να έχουν τη δυνατότητα και άλλοι να μπουν στην αγορά και να συνεργαστούμε. Θα κάνουμε λοιπόν μια σχετική πρόταση από αυτού. Euh, Ευχαριστώ πολύ, Έλγα. Ο κύριος Βόγγελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άλλοι είπαν ότι ο προπολογισμό 2011 θα είναι δύσκολο και δεν υπάρχει εμβολία ότι οι συζητήσει θα είναι δύσκολε και οι συζητήσει για τον προπολογισμό μα του 2011. Το είδαμε λίγο και θα το δούμε και αργότερα όταν θα μιλήσουμε για τον τροποποιημένο προπολογισμό του 2010 γιατί οποτεδήποτε μιλάμε για περισσότερα χρήματα προκύπτουν προβλήματα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να θεσπίσουμε τις προτεραιότητές μας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Για τον προπολογισμό του 2010 που έχει φτιάξει ο κ. Μάγκα υπάρχει το θέμα όπως η ανθρώπινη πόρη, η οργάνωση, περισσότερη και καλύτερη ενημέρωση για τους ευρωβουλευτές. Επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να τονίσουμε την κτηριακή πολιτική, την επικοινωνία και τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ορισμένα επιτέφθησαν, αλλά ορισμένα άλλα ίσως να θεωρούμε πως δεν είναι, ακόμα, δεν είναι πια προτεραιότητες και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια τέτοια συζήτηση το δυνατό συντομότερο. Έχουμε υποχρεωτικέ και μη υποχρεωτικέ δαπάνε, αλλά βασικά αφορά τι επιλογέ που θα κάνουμε για τα πράγματα στα οποία πρέπει να δαπανίσουμε και αυτά που ίσω να μην χρειάζεται να δαπανίσουμε στο μέλλον. Να κάνουμε λοιπόν μια τέτοια δουλειά, να δούμε ποιε είναι οι δυνατότητέ μα για να μπορέσουμε να λάβουμε τι αποφάσει μα με βάση τι προτεραιότητε. Υπάρχουν και άλλα θέματα που νομίζω θα πρέπει να εξετάσουμε, όπως η κτηριακή πολιτική, το αν χρειάζεται να χρηματοδοτήσει η χρηματοδότηση αυτή να είναι σε πιο μόνιμη βάση, γιατί η αιτήσια, ο αιτήσιος προγραμματισμός είναι δύσκολο, καθιστά μάλλον δύσκολη τον προγραμματισμό για αγορές ή συντήρηση κτηρίων. Εγώ νομίζω πως θα πρέπει αυτό να το διαπραγματευτούμε εκ νέου αυτή την συμφωνία κυρίων, γιατί έχω την εντύπωση στο μέλλον ο αριθμός αυτός δεν θα είναι βιώσιμος αν θέλουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο εργασίας του Κοινοβουλίου. Πολλά πράγματα λοιπόν πρέπει να συζητηθούν. Πιο σημαντικό όμως είναι να γίνει αυτή η πρώιμη συζήτηση για τις προτεραιότητες μας. Συζήτηση με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε, ο κύριος Φερνάνδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω την εισηγήτρια και να της πω ότι το ΕΛΚ είναι διαθέσιμο για τους στόχους που απαρίθμησε εν γέννη είναι, και επίσης θεωρεί και επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι η προτεραιότητά μα θα πρέπει να είναι η νομοθετική αριστεία. Εάν δεν έχουμε εξαιρετική νομοθεσία, αυτό θα σημαίνει μεγάλη κόστος για την Ευρώπη και για τους πολίτες της. Και για το στόχο αυτό είναι σημαντικό να υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα ώστε να υλοποιηθεί. Ως εκ τούτου, για ό,τι και αν κάνουμε, θα πρέπει καταρχήν να υπάρχουν τα διαθέσιμα τα μέσα για τους βουλευτές, τις επιτροπές και τις πολιτικές ομάδες. Είναι πήγον να γνωρίζουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Είναι επίγον να γνωρίζουμε τις σταθερές δαπάνες που βρισκομαστε ειναι πηγον Ήδη έχουμε επιμείνει επανειλημμένα για το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και θα ήταν πολύ χρήσιμο σε αυτό το νέο πλαίσιο, με τη νέα δηλαδή συνθήκη, να προχωρήσουμε προς έναν προπολογισμό με μηδενική βάση, όπου η προτεραιότητα για την νομοθετική αριστεία να είναι σαφής. Ανέκαθεν λέγαμε ότι η πολιτική αυτή θα είναι, η κλιμαλεκτηριακή έχει μεγάλη βάρος όσον αφορά τον προπολογισμό. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό το σοφόρτος κάπως να κατανεμηθεί και ίσως και να αναθεωρηθεί, να αναθεωρηθεί αυτή η πολιτική. Ώστε να μην είναι αυτή η προτεραιότητά μας. Τώρα όσον αφορά την συμφωνία που είπαμε, που αποκαλείται μάλλον η Συμφωνία Κυρίων, είναι μια αυτοκυριαρχία, ας πούμε, για το 20%. Θα ήταν σημαντικό να έχουμε ένα μήνυμα, να προσπαθήσουμε να δούμε αν θα μείνουμε και θα επιμείνουμε σε αυτό το 20%. θα πρέπει καταρχήν να περικόψουμε ό,τι δεν είναι απαραίτητο και γι' αυτό είναι σημαντικά τα σταθερά, οι σταθερές δαπάνες και ο προπολογισμό με μηδενική βάση. Να περικόψουμε εκεί που μπορούμε να περικόψουμε στα όσα δεν είναι προτεραιότητες και με στη συνέχεια αφού θα γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε και θα έχουμε παληθεύσει τι χρειαζόμαστε ακριβώς, αν δούμε πως το 20% δεν αρκεί για την προτεραιότητα αυτή που είναι η νομοθετική αριστεία, τότε θα πρέπει να προβλέψουμε και να ξαναδούμε αυτό το ανώτατο όριο του 20%. Να μην είμαστε φανατικοί σε αυτό το θέμα, καθώς επιπλέον Εάν υπάρχει ένα θεσμό στον οποίο ζητείται μεγαλύτερο φόρτο, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό και ακριβώ. Και διότι πάντοτε διατρέχουμε τον κίνδυνο να γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να αναζητήσουμε συνένεση. Πρώτα να δούμε ποια είναι τα περιτά στοιχεία που μπορούμε να αφαιρέσουμε από τον προπολογισμό, πού μπορούμε να εξοικονομήσουμε και μετά αν δεν μπορούμε να εξοικονομήσουμε όσο θα έπρεπε να διαπραγματευτούμε με τα άλλα θεσμικά όργανα και με το Συμβούλιο ώστε να μην υπάρχουν ε, ε, συγκρούσεις ε, διοργανικές για να δούμε ακριβώς τι χρειαζόμαστε για να μπορούμε σωστά να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πόρτας. Εγώ νομίζω πως η συνάδελφος Έλκα Τρούπελ έχει την μεγάλη αρετή ότι έθεσε το, τα πιο δύσκολα θέματα και τα πιο μεγάλα προβλήματα. Όντως είναι αυτά αν ας πούμε στο σημείο που θα συζητήσουμε σε μισή ώρα προβλέπονται 3 εκατομμύρια για 6 μήνες, μπορούμε να βασιστούμε, να υπολογίζουμε στα 26 εκατομμύρια και όχι στα 23 για το 2010. Πέρα από όλα τα άλλα που ανέφερε. Μιλήσαμε για 157 εκατομμύρια ευρώ, ευρώ μιλήσαμε για την αύξηση των ε, διαφόρων δαπανών με βάση την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας και όλα αυτά είναι συμφωνημένα. Το θέμα είναι γύρω στο 4% θα αυξηθεί ο προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Δεν είναι πολύ εύκολα βιώσιμη μια τέτοια αύξηση ανάμεσα στα διάφορα πολιτικά θεσμικά όργανα και γι' αυτό και συμφωνώ ότι θα πρέπει σοβαρά να συζητήσουμε ακόμα μια φορά το θέμα των δαπανών. και να δώσουμε τη δέουσα προσοχή. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο, ένα σημείο το οποίο θα ήθελα οπωσδήποτε να εξετάσουμε. Η συμφωνία η διοργανική που έχουμε λέει ότι στην ουσία κανένα δεν ανακατεύει του λογαριασμούς του αλλονού για κάθε ένα από τα θεσμικά όργανα. Αλλά εγώ πιστεύω πως έχουμε όλοι μα μια ιδέα ότι σε ορισμένου τομεί για την λογική χρήση των μέσων κοινά εν γέννη από τα θεσμικά όργανα τελικά οδηγεί σε μεγάλες ε, σπατάλες. Γι' αυτό θα πρέπει να ξαναδούμε αυτή την συμφωνία. Έτσι ώστε ο καθένα να έχει τους λογαριασμούς του και να φτάνει μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Το πρόβλημα δεν είναι όμως το ποσοστό, το πρόβλημα είναι το σύστημα που έχουμε. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρο το στένος, για να αρχίσουμε να αμφισβητούμε κάποιε παροχέ υπηρεσιών. Δεν μιλάω για όλου, για όλες. σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση κονδυλίων. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε λοιπόν υπόψη γιατί ενώ έχουμε δικαίωμα για συμβολή του βελγικού κράτους στο επόμενο χρόνο, το μεθεπόμενο χρόνο θα έχουμε πάλι να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα και γι' αυτό ίσως θα πρέπει να βρούμε πιο βιώσιμες λύσεις όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες. Σας ευχαριστώ. Έλγα. Ποια είναι η γνώμη σας μετά τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Πρώτα, ευχαριστώ όλους και όλους για τα σχόλια και τις ε, προτάσεις τους. Ο εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος είπε ότι αφενός υπάρχουν λόγοι να εμείνουμε στα 20% αλλά ότι βέβαια δεν είναι και φανατικά υπέρ και ότι στις επόμενες εβδομάδες θα εξετάσουμε το θέμα. Ούτε εγώ θέλω να τηρήσω διαφορετική στάση από αυτήν που μου είπε η Σιδονία. Αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει σπατάλη ή ότι μπορεί να υπάρξει καλύτερη διαχείριση σε ορισμένε υπηρεσίε ή αν μπορούν να γίνουν κάποιε μεταφορέ από εδώ και από εκεί. Ασφαλώ αυτή πρέπει να είναι η προσπάθειά μα να χειριζόμαστε τα χρήματα με τον καλύτερο και πιο υπεύθυνο δυνατό τρόπο. Ταυτόχρονα όμω να μην λησμονούμε, να μην χάνουμε τον στόχο από τα μάτια μας ότι πρέπει να διαμορφώσουμε και τον τρόπο εργασίας μας με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Αυτός πρέπει να είναι επίσης στόχος μας. Για τον λόγο αυτό αναμένω με ιδιαίτερη ανυπομονησία τη συνεργασία μαζί σας για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες και νομίζω ότι αυτό θα είναι σημαντικό και για την πολιτική συζήτηση αλλά και για την καλή διοίκηση του οίκου μας για το πώς θα διαμορφώσουμε τελικά αυτό τον προϋπολογισμό του 2011 αυτό θα είναι κρίσιμο και ως πολιτικό μήνυμα. Νομίζω ότι και όλοι κατανοήσαμε ότι η αντιπαράθεση με το Συμβούλιο Υπουργών στο θέμα αυτό δεν θα είναι βέβαια εύκολη. Ευχαριστούμε, Χελγά. Το είπαμε και στην ψηφοφορία του προϋπολογισμού για το 2010. Το είπαμε και στη συζήτηση για το διορθωτικό προπολογισμό του 2010 μετά από έκθεση του Βλαντιμίρ Μάνικα. Διανύουμε μια χρονιά που θα μας φέρει αντιμέτωπους με ένα δίλημα για όλους τους προϋπολογισμούς και ιδιαίτερα για το δικό μας, το ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Γιατί αφενός ε, η εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας καθιστά αυτή τη χρονιά μια χρονιά που χρειάζεται αύξηση του προπολογισμού για να ανταποκριθούμε στην αύξηση των αρμοδιοτήτων μας. Απ' την άλλη βιώνουμε την χειρότερη οικονομική κρίση με τα πολεμικά. Οπότε και οι εθνικοί προπολογισμοί αλλά και ο κοινοτικό προπολογισμό θα υποστούν σημαντικούς περιορισμούς και έτσι έχουμε αντικρουόμενες πολιτικές απαιτήσεις. Ευχαριστώ, Έλγα, και όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 8, τη γνωμοδότηση που θα καταρτήσει η Επιτροπή μας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γεωσκόπησης με δορυφορικό σύστημα, GMS. Θα δώσω το λόγο στον συντάκτη της γνωμοδότησης, τον κύριο Νταμιά Αμπάντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η θέση σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα με τη δημιουργία μια νέα νομική βάση για το διάστημα και η παρουσίαση των πολιτικών προτεραιοτήτων τη Νέα Επιτροπή, όπω αυτέ εκτέθηκαν από τον πρόεδρο Μπαρόζο, ανάγουν τη διαστημική πολιτική σε ένα από του τομεί κλειδιά για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, πριν ασχοληθούμε με του οικονομικού και δημοσιονομικού περιορισμού και τα δικαιωμένα, α δούμε τα πολιτικά προβλήματα του GMS γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα GMS. Θα έχει απτά αποτελέσματα για τους πολίτες, είτε σε θέματα απασχόλησης, τεχνογνωσίας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Μάλιστα, ε, ο πρόσφατος σεισμός στην ΑΕΤ μας έδειξε πως οι δορυφορικές εικόνες, ιδιαίτερα από το GMS, μας επέτρεψαν να, να προσδιορίσουμε πολύ γρήγορα τις πληγήσεις ζώνες και έχουμε ένα απτό παράδειγμα χρήση τη διαστημική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαστημική πολιτική, βέβαια, ε, σημαίνει και βούληση μια γνήσια βιομηχανική πολιτική ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση συγκεκριμένα προγράμματα και σχέδια. Επίση, έχουμε και θετικέ συνέργειε για άλλου οικονομικού τομεί, όπω οι υπηρεσίε, δημιουργώντα έτσι σημαντικέ ευκαιρίε για την είσοδο στην αγορά ενό μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει όμως να ασχοληθούμε κυρίως με το θέμα της χρηματοδότησης του προγράμματος, ε, εξετάζοντας και την βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη προοπτική. Σε ό,τι αφορά την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, φυσικά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη θέση εφαρμογή του προγράμματος αυτού και η εν λόγω πρόταση προβλέπει την δημιουργία μιας νομικής βάσης που διασφαλίζει τη συνέχεια των προπαρασκευαστικών ενεργειών που θεσπίστηκαν με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρόγραμμα GMS που έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια έχει κινηθεί ως σήμερα στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη που έχει χρηματοδοτηθεί με ποσό 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 2007-2013. Επίση, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο συμμετέχει από την πλευρά του στην ανάπτυξη του προγράμματο με 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε θα ήθελα να σας εξηγήσω το περιεχόμενο της δεύτερης τροπολογίας μου σε αυτό το πλαίσιο, γιατί το σύνολο της χρηματοδότησης στα πλαίσια του 7ου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου για το GMS ανταποκρίνεται σε 43 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ που είναι στα πλαίσια του διαστήματος, 43 εκατομμύρια ευρώ και εκεί θα πρέπει να προσθέσουμε 43 στα 2009 και τα 166 εκατομμύρια ευρώ που ήταν κονδύλια από δημοσιονομικές γραμμές που υπήρχαν ήδη για το GMS στα πλαίσια του 7ου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου και έχουν ήδη προβλεφθεί για τη χρησιμοποίηση και τη συνέχιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος. Η φάση ανάπτυξη και έρευνα ε, φτάνει στο τέλος και από το 2011 θα περάσουμε στην πιο επιχειρησιακή φάση του προγράμματος. Γι' αυτό και θα πρέπει να βρούμε νέες πηγές κοινοτική χρηματοδότησης. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα επιπλέον κονδύλιο, 107 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ορισμένες επιχειρησιακές αποστολές του προγράμματος. Υπάρχουν πολλές οικονομικές δυσκολίες στο πρόγραμμα αυτό. Η κατηγορία 1α, όπως είπαμε και στην προηγούμενη συζήτηση, υφίσταται τεράστιες πιέσεις και έχει περιορισμένα κονδύλια και βλέποντας ε, την εξέλιξη μεταξύ 2011 και 2013 βλέπουμε 10 εκατομμύρια το 2011, 41 το 2012 και 56 το 2013. Κάτι που αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επιπλέον κόστος για έναν ήδη υπερφορτωμένο τομέα. Επίσης, ε, πρέπει να προσδιοριστούν και οι ακάλυπτες ανάγκες που δεν έλεγχαν υπόψη στο πολιετές πρόγραμμα πλαίσιο. Για παράδειγμα, το διαστημικό σκέλος του προγράμματος, γιατί τρία είναι τα σκέλη του προγράμματος. Το θεσμικό και το διαστημικό, αλλά και το, το σκέλος των υπηρεσιών. Σε, σε ό,τι αφορά το διαστημικό σκέλος, οι εμπειρογνώμονε επισήμαναν ότι έχουν μείνει αχρηματοδότητε κάποιες ε, ε, επιχειρήσεις με, σε ύψο 200 ε, με 300 εκατομμύρια ευρώ όπως επισημαίνει και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Οπότε για να δεσμευτούμε και βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να καθορίσουμε μια δημοσιονομική πολιτική σαφή για το πρόγραμμα μετά το 2013. Χρειαζόμαστε ένα πλήρω ανεπτυγμένο πρόγραμμα GMS στα πλαίσια του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, γιατί όλοι συμφωνούμε ότι οι ανάγκε χρηματοδότηση του προγράμματο είναι μεγαλύτερε από τι πιστώσει που διατίθενται σήμερα. Αν θέλουμε ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε τις επιχειρήσεις του δορυφόρου Sentinel-Α, να τροφοδοτήσουμε το Sentinel v και να ε, εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό και τη χρηματοδότηση του Sentinel Γ. Αυτά λένε και τροπολογίες 3 ε, και 4. Κυρίως οι 4. Αυτό προς το βραχυπρόθεσμο αλλά έχουμε και τα θέματα τα πιο μακροπρόθεσμα και τι επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικές. Το 2010 έχουμε καταρχήν την ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020, την ενδιάμεση αναθεώρηση του 7ου ερευνητικού προγράμματο πλαισίου και την ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου που περιλαμβάνει κυρίω τη χρηματοδότηση των νέων πολιτικών που προβλέπονται από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Μην ξεχνάτε και τη χρήση του μέσου ευελιξία, καθώ και τη χρήση τη νομοθετική ευελιξία όπως προβλέπει το άρθρο 37 της Διοργανικής Συμφωνίας. Κάτι που, είναι σημαντικό, κάτι που αποτελεί σημαντικό εργαλείο. Και θα ήθελα εδώ να παταθώ στο Συμβούλιο που πολύ συχνά ξεχνάει αυτά τα μέσα που είναι πολύ χρήσιμα και γι' αυτό το επισημαίνω στην τροπολογία 3. Οπότε είναι άρρηκτα συνδεδεμένα το βραχυπρόθεσμο με το μέσο και μακροπρόθεσμο σκέλος. Για την περίοδο 2014-2020 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για την περίοδο την επιχειρησιακή του 2011-2013. Μετά από διαβουλεύσεις που είχαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και το, τη βιομηχανία, είδαμε ότι κάποια θέματα αφορούν κυρίως την ιδιοκτησία των υποδομών, την ε, πολιτική διαχείριση των δεδομένων, πολιτική επιπτώσεων του διαστημικού προγράμματος, αλλά και θέματα διεθνού συνεργασία με τις τρίτες χώρες και πολιτική προμηθειών για τη διαστημική υποδομή του GMS. Μολώνοντα η συνεργασία μεταξύ Επιτροπή και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματο λειτουργήσε κατά τη φάση τη έρευνα και ανάπτυξη, κρίνεται αναγκαία κατά την επιχειρησιακή φάση να διευρυνθεί η διαδικασία αυτή διαβούλευση. Με αυτή την έννοια προτείνουμε την δημιουργία ενός Συμβουλίου των Εταίρων, το οποίο οι αρμοδιότητε θα είναι συμπληρωματική επιτροπή GMS που προβλέπεται στην πρόταση κανονισμού. Και στόχο μας είναι να συμπληρώσουμε αυτή την επιτροπή GMS με μια υπάρχουσα δομή που έχει όμως προσωρινό χαρακτήρα, με ελάχιστο κόστος, σχεδόν μηδενικό, προκειμένου να υιοθετήσουμε μια δημοσιονομική συντονισμένη στρατηγική σε πολλαπλά επίπεδα. Αυτή η δημιουργία του Συμβουλίου Εταίρων δεν είναι δική μου επινόηση τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν ομόφωνα συμφωνήσει στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα του Δεκεμβρίου του 2008 να ιδρύσουν αυτό το Συμβούλιο των Εταίρων με στόχο να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την κατάρτιση μέσω και μακροπρόθεσμης στρατηγική. Γι' αυτό και προτείνω ένα άρθρο στην τροπολογία 5 για τη σύσταση αυτού του Συμβουλίου των εταίρων και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μία μέσο και μακροπρόθεσμη στρατηγική χρηματοδότηση του προγράμματος μέχρι το Δεκέμβριο του 2010. Στο τελευταίο αυτό άρθρο περιλαμβάνονται και κάποια ενδιάμεσα μέτρα διοίκησης και διαχείρισης. Ήδη υπάρχει αυτό το Συμβούλιο των Εταίρων που, επαναλαμβάνω, λειτουργεί προσωρινά. Καλό θα ήταν να το θεσμοθετήσουμε πιο επίσημα και να το εφοδιάσουμε με επιπλέον μέσα, μέσω μιας αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό του προγράμματος GMS, κάτι που απαιτεί δέσμευση τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και των κρατών μελών. Και έχουμε μια τεράστια ευκαιρία και μια πρόκληση όμως, και μάλιστα όλα αυτά συνάδουν με τις προθέσεις και τις προσδοκίες των εισηγητών του προπολογισμού του 2011. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο Γκέραν Φέρμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ παρεμβαίνω αντικαθιστώντας την κυρία Χέρτζοκ, την σκιά ηγήτρια που πρέπει να βρίσκεται σε μια άλλη συνεδρίαση. Ω ταμέα ε, τη ε, σοσιαλιστική ομάδα, ε, έχω μια ερώτηση. Είναι προτεραιότητα, αναφίβολα. Είναι σημαντικό από βιομηχανική άποψη, είναι πολύ σημαντική τεχνολογία και από περιβαλλοντική άποψη και από άποψη κλιματικών αλλαγών, αλλά δεν έχουμε καταλάβει τη χρηματοδότηση. Εδώ υπάρχουν ένα σωρό νούμερα. Από ό,τι κατάλαβα υπάρχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Οργανισμό Διαστήματος, χρηματοδότηση από δύο διαφορετικά σημεία του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη και από πάνω χρειάζονται και 107 επιπλέον εκατομμύρια ευρώ. κατάλαβα καλά. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε πώς από αυτά είναι για το 2011 από, τις διάφορες αυτές, από τα διάφορα αυτά κονδύλια. Και έπειτα ε, υπάρχουν και άλλοι πόροι όπως η ε, ιδιωτικές, ε, η ιδιωτική συνεργασία για παράδειγμα. Δεν έχουμε την πλήρη εικόνα για το 2011 και δεν ξέρω αν είναι η Επιτροπή που πρέπει να το διευκρινίσει ή ποιος πώ είναι οργανωμένα τα πράγματα ή αν πρέπει ο εισηγητή να τα διευκρινίσει. Δεν έχουμε πάντω πλήρη εικόνα και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όλα τα άλλα κομμάτια τη χρηματοδότηση εμπίπτουν κάτω από το ανώτατο όριο του δημοσιονομικού πλαισίου. Δηλαδή, μόνο τα 107 εκατομμύρια, από τα οποία 10 είναι για την επόμενη χρονιά, είναι αυτό το μόνο πρόβλημα από την άποψη του ανώτατου ορίου τη οροφή. αν είναι μόνο 107 εκατομμύρια, εντάξει, δεν είναι και μικρό το ποσό βέβαια. Αν δούμε τα προβλήματα που έχουμε με την κατηγορία 1α, είναι πραγματικά προβληματική. Ήδη για το 2011 πιστεύω λοιπόν πως η Κομισιόν ή ο εισηγητής θα πρέπει αυτό να μας το αποσαφηνίσουν. Και λόγω του προβλήματος με το δημοσιονομικό πλαίσιο θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή για την τροπολογία 1 όπου θίγει αυτό το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω πως θα πρέπει να είμαστε ίσως ακόμη πιο σαφείς από ότι είναι ο ίδιος, γιατί λέει ότι είναι σημαντικό λέει πω θα είναι συμβατό με το ενοροφή μόνο από τη στιγμή που όλοι οι διαθέσιμοι μηχανισμοί που ισχύουν σύμφωνα με τη Διοργανική Συμφωνία και αναφέρει τα σημεία 20 21 μέχρι 23 και 37 ε, χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει να είναι λοιπόν σαφές. Είναι αυτό απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει αναθεώρηση του, της γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε. Κάπως λοιπόν να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Κάποιος μπορεί να μας διαφωτίσει για την πλήρη εικόνα όσον αφορά την χρηματοδότηση για το 2011. Ευχαριστώ, Γκέρχαν. Ο κύριος Χάντλουντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, συνάδελφοι, για την εξαιρετική σας έκθεση. Ο και ο Γιώργος έδειξαν το ίδιο είδου ερωτήσεις όπως και αυτές που θέλω εγώ να θέσω γιατί μόνιμος, ε, είμαι μόνιμος συζητητής για την έρευνα για φέτος και έχω κάποιες ερωτήσεις για τα ίδια θέματα. Καταρχήν με ανησυχεί ιδιαίτερα το, το κομμάτι της χρηματοδότησης γιατί όπως ίσως γνωρίζετε και όπως αναφέρθηκε το πρόγραμμα παρατήρηση τη γης χρηματοδοτείται, ε, χρηματοδοτείται από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Μιλάμε για 107 επιπλέον εκατομμύρια και επειδή ξέρουμε την κατάσταση με την κατηγορία 1α, θα ήθελα να δω πώς η Κομισιόν σκοπεύει να το χρηματοδοτήσει. Ο εισηγητής λέει πως σκοπεύει να το χρηματοδοτήσει ανεξάρτητα από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Από τη μια πλευρά είναι καλό, από την άλλη πλευρά ξέρουμε πως μπορεί να μην είναι δυνατόν να βρεθούν τα χρήματα. Και, και ταυτόχρονα η νομική βάση αφορά το πρόγραμμα γεωσκόπησης και ε, μπορεί να υπάρξει και η πρόθεση από πλευρά τη Κομισιόν να χρηματοδοτήσει τα 107 εκατομμύρια από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Και, αυτό δεν θα μου άρεσε καθόλου γιατί προχωράμε στο λειτουργικό, στη λειτουργική φάση. Γι' αυτό και δεν ξέρω αν θα ήταν σκόπιμο να χρηματοδοτηθούν από αυτό. Και έπειτα η Κομισιόν ζητά ακόμα 43 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή 150 εκατομμύρια ακόμα, πάνω από τα 106 που είχαμε, 160 που είχαμε πριν. Ε, δηλαδή 310 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Ε, πολλά χρήματα. Θα ήταν σημαντικό λοιπόν όλα αυτά να επαληθευτούν. Προπαρασκευαστικές τώρα δράσεις για το 2011. Να πάμε και στο 11 ε, και εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ποια ποσά θα θεωρηθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Να σας θυμίσω επίσης ότι αν υπάρχουν 150 εκατομμύρια ευρώ Επιπλέον, αυτό σαφώ δείχνει ότι πρέπει να γίνει μια ενδιάμεση αναθεώρηση του 7ου προγράμματο πλαισίου. Ε, και αν όχι, θα ήθελα να ξέρω πού θα τα βρούμε αυτά τα χρήματα. Χρειάζονται διευκρινήσει λοιπόν, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την καλή έκθεση έχετε τονίσει πολλές από τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ. Ο Χάιμερ Μπέγκε. Σας ευχαριστώ. Η παρέμβαση του κυρίου Έντλουντ με οδηγεί να παρέμβω και να θέσω μια ερώτηση στην Κομισιόν. Όχι μόνο για την έρευνα έχουμε το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά για όλα τα πολιετή προγράμματα έχουμε μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Το 2010 για όλα τα πολιετή προγράμματα προβλέπεται αναθεώρηση. Είναι τμήμα της, της πολιτικής συμφωνίας που έχουμε συνάψει στο πλαίσιο της ε, συναπόφασης και της διαβούλευσης. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω, ίσως όχι άμεσα σήμερα, αλλά στις επόμενες μέρες η Κομισιόν θα πρέπει να μας κάνει μια ανακοίνωση για αυτά τα θέματα για το σε ποιο βαθμό δηλαδή μέσα σε κάθε μία από τις αρμόδιες ε, γενικές διευθύνσεις η ενδιάμεση αξιολόγηση για το δημοσιονομικό και τεχνικό επίπεδο θα γίνει. Δηλαδή πότε θα ξεκινήσει αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση και πότε σκοπεύει να ασχοληθεί με το θέμα η Κομισιόν ή νομίζετε ότι θα την κάνει μόνο του το Κοινοβούλιο. merci, Ευχαριστώ, Ράιμερ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμη σχετική επιτροπή. Ναι. Νομικός ναι, αλλά διοικητικός ελάχιστα. Και πολιτικό είναι κάπως μετέωρη. Πρέπει το Κοινοβούλιο τη σοφία του να την επικυρώσει την επόμενη εβδομάδα. Οπότε δεν μπορούμε να θέσουμε πολιτικά ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Μπορούμε όμως να θέσουμε τεχνικά ζητήματα. Όπως πρότεινε και ο συγητής μας ε, και μετά συμφώνησαν και ο Γκέραν και ο Ράιμερ, αν δεν λάβουμε κάποιες διευκρινήσεις τις επόμενες εβδομάδες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε όλες τις γνωμοδοτήσεις που θα χορηγούμε θα λέμε το ίδιο, ότι είναι συναρπαστικό με το πρόγραμμα, αλλά το ταμείο είναι μείον. Είμαστε υπέρ του προγράμματος υπό τον όρο της αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών. Δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Και είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση και δεν μας περιπεί Υπάρχουν και πολλές συγκεκριμένες ερωτήσεις για τα ποσά και τις δημοσιονομικές γραμμές που εμπλέκονται ή τους άλλους εταίρους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ή κάποιες ε, συμπράξεις ιδιωτικού, ιδιωτικού δικαίου ή ιδιωτικών φορέων. Και τι τμήμα θα εφοδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον προπολογισμό του 2011. Δεν ξέρω, για τα σημεία αυτά θα μπορούσαν να μας ε, δώσουν κάποιες απαντήσεις εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ή να ζητήσουμε από τον εισηγητή μας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις επαφές που θα έχει μαζί της να περιμένουμε ένα γραπτό δελτίο με τις διευκρινήσεις αυτές ώστε να είμαστε ενημερωμένοι πριν ψηφίσουμε. Γιατί μην ξεχνάτε την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών που λύγει την επόμενη εβδομάδα στις 2 Φεβρουαρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει στις 4 Μαρτίου. Δεν ε, επήγει το θέμα αλλά χρειαζόμαστε αυτέ τι διευκρινήσει πριν να αποφασίσουμε. Κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο, ο κύριο Γενικό Διευθυντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το πρώτο σα σχόλιο θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα υποβάλει προτάσει αν δεν μπορεί να τι χρηματοδοτήσει κιόλα. Φυσικά υποβάλλουμε προτάσει χρηματοδότηση μπορεί να δυσαρεστούν ορισμένου. αλλά θα αποφασίσει γι' αυτό η αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή. Πάντως υποβάλλουμε προτάσεις με τρόπους χρηματοδότησης. Και αυτό ισχύει και για το πρόγραμμα GMS. Σε ό,τι αφορά τις διευκρινήσεις που ζητήσατε, έχω κάποια στοιχεία, αλλά πολύ φοβούμαι ότι θα είναι βαρετό και περίπλοκο να σας τα εξηγήσω. Αφήστε που μπορεί να παρεξηγηθούν και όλα. Θα σας μοιράσω πάντως ένα δελτίο για να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ της χρηματοδότησης των εργασιών, των δραστηριών και των επιχειρησιακών αποστολών του GMS. Τα 107 δηλαδή εκατομμύρια ευρώ. Προτιμώ να σας μοιράσω αυτό το δημοσιονομικό δελτίο. Για τα 107 εκατομμύρια πάντως δεν ξεπερνούμε το περιθώριο και για τα 107 εκατομμύρια, 22 εκατομμύρια είναι ανακατανομή που προέρχονται από το πρόγραμμα ΣΥΠ και 85 εκατομμύρια από το περιθώριο. Οπότε θα ήθελα να σας καθησυχάσω ότι δεν θα το ξεπεράσουμε το περιθώριο. Πάντως θα σας παράσχουμε ένα πλήρες δημοσιονομικό δελτίο, μην ανησυχείτε. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Διευθυντά. Όντως, στον προϋπολογισμό το πιο βαρετό πράγμα είναι τα ποσά, η αριθμία, αλλά είναι και το πιο σημαντικό σε έναν προϋπολογισμό. Οπότε θα πρέπει να προβλέψουμε άλλες ευκαιρίες για χαμόγελα. Κύριε Σιγητά, ποια είναι η γνώμη που διαμορφώσετε μετά τη συζήτηση. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση με τις χρήσιμες και εύστοχες παρατηρήσεις τους και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διευκρίνηση ως προς τα 107 εκατομμύρια ευρώ. Δύο είναι πάντως οι φάσεις του προγράμματος. Υπάρχει η ερευνητική φάση και η φάση ανάπτυξης που αντιστοιχούν στα 209 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή τα 166 εκατομμύρια που ήταν σε προηγούμενες δημοσιονομικές γραμμές, είναι τα 43 εκατομμύρια που προέρχονται από τη γραμμή για το διάστημα. Αυτά για την έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτή είναι η μία φάση και η άλλη φάση είναι η επιχειρησιακή, όπως εξήγησε και ο Γενικός Διευθυντής, που θα τεθεί σε ισχύ από το 2011 και μετά. Και ακριβώ επειδή υπάρχει και η επιχειρησιακή φάση, θα πρέπει να προσθέσουμε επιπλέον 107 εκατομμύρια ευρώ. Και για το 2011 θα έχουμε 10 εκατομμύρια για την επιχειρησιακή φάση, 41 εκατομμύρια το 2012 και 56 εκατομμύρια το 2013. Αυτά για την επιχειρησιακή φάση. Πάντως, ε, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος είχαμε 1,6 εκατομμύρια μέχρι το 2006 και για την περίοδο 2007-2013 1,2 δισεκατομμύρια. Και σας είπα, τα 209 βγαίνουν από τα 166 συν 43. Θα υπάρξει συνέχιση και της ε, ερευνητικής και αναπτυξιακής φάσης. Γι' αυτό και έχουν απομείνει κάποια κονδύλια στην ε, ερευνητική και αναπτυξιακή φάση. Αλλά χρειαζόμαστε ένα συνοπτικό δελτίο για να έχουμε όλα τα κονδύλια μαζί και να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να χρηματοδοτήσουμε αυτή την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Θα πρέπει όλα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία και αυτά τα ποσά να τα κατατάξετε σε ένα δημοσιονομικό δελτίο, ώστε όλοι να μπορέσουν να ενημερωθούν και να ψηφίσουν ε, έχοντας γνώση. 2 Φεβρουαρίου λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες, 4 Μαρτίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και 17-18 Μαρτίου θα ψηφίσει αρμόδια κατουσία Επιτροπή που είναι η Επιτροπή Βιομηχανίας, Ήτρε. Τώρα για το σημείο 7 είχα υποσχεθεί στον Ζαλουκ Τεάνο το σημείο 7 θα το εξετάζαμε από τις 5 και μετά. Είναι 5 και 10, οπότε Ζαλίκ έχετε το λόγο για ένα θέμα στο οποίο θα χρειαστεί η πλούσια πολιτική σας πείρα και είναι ο τρόπος υπολογισμού του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος. Εμείς ε, <laughs> το... Εμείς ε, μαζί με το Νεπάλ είμαστε αυτοί που υπολογίζουμε το... την ακαθάριστη εθνική ευτυχία. Μόνο εμείς και το Νεπάλ, η Γαλλία και το Νεπάλ υπολογίζουν ε, αυτό το στοιχείο στο καθάριστο εθνικό προϊόν. Αν περιμένουμε να συμπεριλάβουμε στο ΑΕΠ και το, την καθάριστη εθνική ευτυχία, θα περιμένουμε άλλα 10 χρόνια. Εδώ 10 χρόνια περιμένουμε για το ΑΕΠ. Όπως είπα, δεν είναι καινούργιο αυτό το θέμα, γιατί η νομική βάση προτάθηκε το 1998 και πρόκειται για τον τρόπο υπολογισμού του καθάριστου εθνικού εισοδήματος με βάση το οποίο υπολογίζουμε ένα τμήμα των ιδίων πόρων της Ένωσης και εκεί θα προσθέσουμε και ένα τμήμα των υπηρεσιών που προσφέρουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Είχαμε λοιπόν τη νομική βάση το 1998 που έπρεπε να εφαρμοστεί το 2005 αλλά ε, είχαμε προβλέψει μια δοκιμαστική περίοδο για να δούμε τι επιπτώσεις θα είχε και αν θα προκαλούσε αλλαγή άνω του 1% στον προσδιορισμό του καθάριστου εθνικού εισοδήματο. Πέρασε αυτή η δοκιμαστική περίοδος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμαστικής περίοδου είναι επαρκή και προτείνει τη συμπερίληψη αυτού του στοιχείου στον προσδιορισμό του καθάριστου εθνικού εισοδήματο. Μέχρι εδώ ουδέν πρόβλημα και μπορούμε να συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι αρκετά λογική η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί προτείνει τη συμπερίληψη αυτού του στοιχείου την 1η του 2005 γιατί η νομική βάση ανάγεται στο 1998 με πρώτη χρονιά εφαρμογής το 2005. Βέβαια, η διαδικασία αυτή προϋποθέτει ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου με σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Στο Συμβούλιο υπάρχει συμφωνία για το θέμα αυτό, αλλά υπάρχει μία επιφύλαξη ότι αφορά την αναδρομική ισχύ του υπολογισμού. Και από επαφές που είχαμε, γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει να τεθεί σε ισχύ αυτός ο νέος υπολογισμός από το 2010. Πάντως το θέμα κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο σημαντικό για να αρχίσουμε καυγάδες και να διεκδικήσουμε την αναδρομική ισχύ από το 2005, που ούτως ή άλλως και αυτή μπορεί να αφισβητηθεί. Γι' αυτό προτείνω να δεχτούμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί παραλαμβάνω και για το Συμβούλιο υπάρχει συνένεση για εφαρμογή από την 1η Πρώτου 2010. Ας ευθυγραμμιστούμε λοιπόν με το Συμβούλιο και ας μην έχουμε αντιπαράθεση εμένοντας την αναδρομική ίσχυ. Θαυμάσια, Ζανλουκ. Ο Γκέρον. Είχα μια απορία για την λογική αυτή τη απόφαση και για την νομική βάση. Γιατί εφόσον πρόκειται για απόφαση, είναι, θέλει επικύρωση. Αν πρόκειται για εφαρμοστική απόφαση για του πόρου, χρειάζεται μόνο συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είναι απλώ στατιστικό ζήτημα, τότε είναι συναπόφαση, δεν είναι. Οπότε θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι είδου απόφαση είναι αυτή. Κοιτάξτε, ε, είχαμε μια συζήτηση με τις, ε, την νομική υπηρεσία και από ό,τι φαίνεται συμφωνούν όλοι ότι είναι διαδικασία συγκατάθεσης ομοφωνία στην Επιτροπή και ε, συμβουλευτική γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Γιατί είναι πιο στατιστικό το θέμα. πάση περιπτώσει δεν είναι ένα καλό θέμα για να κάνουμε αυτόν τον αγώνα το διαδικαστικό που πρέπει να κάνουμε. Αλλά νομίζω πως δεν, είναι, δεν προσφέρεται αυτό το θέμα. Καλύτερα να ακολουθήσουμε την προδιαδικασία που προτείνει η Κομισιόν. Είναι πιο στατιστική προσέγγιση. Δεν αφορά ε, πραγματικά τους πόρους. Merci de cette précision. Ευχαριστούμε για αυτή τη διευκρίνηση. Είναι μια απόφαση που θεωρούμε ότι εμπίπτει λοιπόν στην στατιστική και άρα στην νομική βάση της στατιστικής και όχι στους ίδιους πόρους. Νομίζω πως η πρόταση του εισηγητή είναι μια λογική πρόταση, εκτός και αν θέλει κανείς να αγωνιστεί για αναθεώρηση με βάση αυτό το νέο, το νέο ορισμό του ΑΕΠ για να υπολογίσουμε την συμβολή των κρατών μελών από το 2005 αλλά πιστεύω πως όπως και συγκεκριτής είναι καλύτερα να το εφαρμόσουμε με βά... από αρχής γενομένης από το 2010 σύμφωνα με τα όσα γίνονται και στο Συμβουλίο. Από ό,τι κατάλαβα είναι επίγον το θέμα. Γιατί η Κομισιόν θέλει να ξέρει από ποιες βάσεις θα επεξεργαστεί το σχέδιο προπολογισμού. Η Γιούτα. Ευχαριστώ. Λέω σύντομα για να μην υπάρξει καμία παρανόηση, αν και ίσως ήταν και θέμα μετάφρασης όταν μιλούσε ο Ζαν δεν πρόκειται για καθαρή στατιστική διότι αλλάζει η βάση υπολογισμού εφού η βάση υπολογισμού περιλαμβάνει περισσότερα από ό,τι πριν άρα δεν πρόκειται για καθαρή στατιστική διότι αλλιώ πραγματικά θα μπαίναμε σε συναπόφαση και θα έπρεπε να ανοίξουμε ολόκληρο το θέμα πάλι όλα αυτά τα έχουμε ξανακάνει ορισμένοι από εσά θα τα θυμούνται αν και είναι κάπω παλαιότερα αλλά και εδώ δεν μας προχωράει καθόλου. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι και η Κομισιόν θα το επιβεβαιώσει. Η Κομισιόν θέλει αναδρομική, αναδρομικό υπολογισμό, διότι τότε αυτά θα σημάνουν παραπάνω χρήματα για τον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Και νομίζω βέβαια ότι και γι' αυτό το λόγο το Συμβούλιο Υπουργών επιμένει ώστε να τεθεί σε εφαρμογή του το, από το 2010. Νομίζω ότι εν προκειμένου δεν θα κερδίσουμε και όπως είπε ο Ζων Λουκ δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να αγωνιστούμε μάταια εάν δεν πρόκειται να επιτύχουμε. Πάντως όπως είπα δεν πρόκειται για την καθαρή στατιστική. Ναι βεβαίω, οι συνέπειες είναι εξάλλου σημαντικές. Μάλιστα. Ο Ζαν Λίκ μας έκανε μια πρόταση. Οι προθεσμοί για τις τροπολογίες είναι 4 Φεβρουαρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμού την επόμενη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα και την ψηφοφορία το Μάρτιο. Στην Ολομέλεια για να είμαστε εντάξει και απέναντι στην Κομισιόν όσον αφορά τα χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, πάει το 7, μπορούμε να περάσουμε στο 10. Γιούτα αντικαθιστά την Edith ΕΡΤΣΟΚ. Α, όχι, συγγνώμη. Ναι. Ναι, ναι, σωστά τα λέω. Λοιπόν, σε σχέση με την διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης. Χάουκ. Υποψιάζομαι ότι ο δισταγμός του Προεδρού οφείλεται στο ότι στην ημερήσια διάταξη αναγράφεται το όνομα Ερτσόκ για, ε, ως εισηγήτρια για τη γνωμοδότησή μας αυτή για αυτή τη νέα αρχή Γαλιλαίο διότι η Edith είναι η διαρκής εισηγήτριά μας για τα θέματα του Γαλιλαίου ωστόσο τούτο το θέμα είναι θέμα για εκείνους που έχουν σχέση για μένα δηλαδή, που έχω σχέση με τους οργανισμούς, εφόσον εντάσσεται σε θέματα οργανισμών. Λέω λοιπόν από την αρχή ότι πρόκειται να υπάρξει έγγραφο την επόμενη εβδομάδα και ναι, ναι, μάλλον την επόμενη εβδομάδα πάντως και θα έχουμε το έγγραφο διαθέσιμο για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών αλλά υπενθυμίζω ότι όταν ο Γαλιλαίος ήταν ακόμα σχέδιο κοινοπραξίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είχαμε αποφασίσει ότι θα δημιουργηθεί μια αρχή ανεξάρτητη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα διαχειρίζεται ορισμένα πράγματα του προγράμματος αυτού και θα τα αξιολογεί. Τώρα ο Γαλιλαίος διαλύθηκε ως κοινοβραξία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και είναι πια καθαρά ευρωπαϊκό έργο. Δεν έχει λοιπόν καμία αξία αυτή η ανεξάρτητη αρχή. Οι χώρες μέλη ούτε επέμειναν άλλωστε να ιδρυθεί εν τέλει Και η Κομισιόν λέει και δικαίω. λέει και δικαίω. ότι δεν θα είναι πλέον ανεξάρτητη. Η Κομισιόν λοιπόν Θα θυμάστε ότι είχαμε ζητήσει κατά επανάληψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προηγούμενη θητεία να μας υποβάλει σχέδιο τροποποιημένης διάρθρωσης για την αρχή του Γαλιλαίου, το οποίο έπραξε τώρα η Κομισιόν. Και στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε το θέμα στη βάση ενός εγγράφου. και εφόσον είναι απαραίτητο θα υποβάλουμε τροπολογίες σε σχέση με τον οργανισμό. Αυτά σχετικά με το γιατί τώρα καλούμαστε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Κανείς δεν ζητεί το λόγο. Καλώς λοιπόν, ευχαριστώ Γιούτα. Όντως, Αντικείμενο της έκθεσης θα είναι η προσαρμογή του καταστατικού και των στόχων του οργανισμού για την έναρξη λειτουργίας του Γαλιλαίου και για τη διαχείρισή του ε, έγιναν μακρές διαπραγματεύσεις μετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της προηγούμενης Επιτροπής Προϋπολογισμών κατέστη εν τέλει απολύτως ευρωπαϊκό έργο. Πρόκειται ωστόσο για το πρώτο βιομηχανικό project κοινοτική ευρωπαϊκής πρωτοβουλία και βασανιστήκαμε πολύ μέχρι να βρούμε τη σωστή φόρμουλα που είναι η φόρμουλα οργανισμού που βέβαια πρέπει ακόμη να διευκρινιστεί και να βελτιωθεί. Η Επιτροπή Ήτρε που είναι αρμόδια επί της ουσίας, θα ψηφίσει στις 4 Τρίτου. Άρα στην επόμενη συνεδρίασή μας θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εγκρίνουμε τη γνωμοδότηση της Γιούτα. Φτάνω στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διαταξής μας, του υπαριθμό 9, του Ράιμερ Μπέγκε, ο οποίος θα μας παρουσιάσει έναν αριθμό φακέλων για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν στις 22 Ιανουαρίου κατέθεσε τρεις προτάσεις για την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, τρεις χωριστές προτάσεις, ακολουθώντας και την αξίωση της Επιτροπής Προπολισμών να γίνονται αυτά τα πράγματα χωριστά και χαιρετίζω την κίνησή της αυτή και από όσο γνωρίζω εξετάζονται και βρίσκονται στον αγωγό προς εμάς άλλα 15 τέτοια σχέδια. Η Επιτροπή Απασχόλησης θα γνωμοδοτήσει ήδη αυτή την εβδομάδα στις 27. Στην επόμενη συνεδρίασή μας θα επανέλθουμε στα σχόλια της Επιτροπής Απασχόλησης με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Άλλο ένα θέμα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Όπως είπα έχουμε τρεις ξεχωριστές προτάσεις, δύο από τη Λιθουανία, αφενός για τον οικοδομικό κλάδο και απώλεια θέσεις απασχόλησης Και τέλος τρίτη από την ε, Ομοσπονδιακή Γερμανία, την αυτοκίνητομηχανία δηλαδή, ένα αυτοκίνητο το οποίο πρόκειται και ένα μοντέλο το οποίο είχε παρουσιαστεί πριν από πολλά χρόνια και ήταν ήδη πολύ επιτυχημένο. Να λοιπόν οι αλλαγές που προκύπτουν. Οι αιτήσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποικίλουν χρονικά από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 23 Ενάτου και η ενδιάμεση κάποια στιγμή τον Αύγουστο. Βλέπω ότι είναι παρόντες και οι πρόσωποι της Κομισιόν. Θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο. Βλέποντας ότι η πρώτη αίτηση από τη Λιθουανία για κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων αναφέρεται σε 600 φυγωμένους οι οποίοι ζητούν υποστήριξη σε έναν αριθμό 480 από το Ταμείο παρόλη την διευκόλυνση των διαδικασιών που είχαμε εγκρίνει προμηνών υπήρξε εδώ εφαρμογή της ρήτρας εξαιρέσεως διότι οι θυγόμενοι εργαζόμενοι εφήγησαν σε δύο φάσεις και 500 εργαζόμενοι δεν φτάνουν στους 500 εργαζόμενους και 4 μήνες κτλ. Για το άλλο όμως, εδώ στο 2C μπορεί να θεωρηθεί παραδεκτή η παρέμβαση του Ταμείου έστω και αν δεν πληρούνται απολύτως οι προποθέσει, διότι οι απολύσεις αυτές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Και η Λιθουανία τονίζει ότι ήδη στην συγκεκριμένη περιφέρεια υπήρξαν παρόμοιες εξελίξεις στην υφαντουρική βιομηχανία, τις οποίες υπεστήριξε, τους θυγωμένους δηλαδή, το Ταμείο. Άρα θεωρώ ορθό ότι γίνεται εφαρμογή της ρήτρα εξαίρεσης ναι. ένα ποσό περίπου 258.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά την πρώτη περίπτωση, 651 εργαζόμενοι, 480 υποτίθεται ότι θα πρέπει να μπορούν να υποστηριχθούν. Στο δεύτερο, κλάδος της οικοδομής, όλα αυτά στο συμπληρωματικό ντοσχέ σημειώνω εδώ ότι αφενός ζητείται εφαρμογή του 2Β, 1612 εργαζόμενοι, σε πάνω από 100 επιχειρήσεις, από τους οποίους ζητείται υποστήριξη μόνο για 806, δηλαδή αφενός μεγάλα νούμερα, αφετέρου όμως ζητεί υποστήριξη μονάχα του ημίσεως. Αν μπορεί η Κομισιόν να εξηγήσει από πού προκύπτουν οι αριθμοί αυτοί και τι γίνεται με τους υπόλοιπους 800. Κάπου μπόρεσαν να απασχοληθούν. Εν πάση περιπτώσει πώς υπάρχει τέτοια μεγάλη διαφορά. Και στη δεύτερη αυτή περίπτωση από τη Λιθουανία είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και παρόλο το μεγάλο αριθμό των επιχειρήσεων έφτασε στις 23 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τον επεξεργάστηκαν την την αίτηση αυτή δύο μήνες ταχύτερα από την πρώτη. Εδώ ζητώ πάλι κάποια εξήγηση. Και τώρα για το Κάμεν στη Γερμανία, δύο επιχειρήσεις που θίγονται από το ίδιο πρόβλημα με 2.500 περίπου εργαζόμενους δύο επιχειρήσεις με συνολικό ύψος αποζημιώσεων 6,2 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να πληρούνται οι άλλες προϋποθέσεις αλλά αναμένεται και η λεπτομερέστερη εξέταση από πλευρά Επιτροπή Απασχολήσεω. Άλλωστε και εγώ τα έγγραφα τα έλαβα μόλι σήμερα το πρωί. Θα ήταν καλό πάντω να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτέ τι πρώτε ερωτήσει. Ευχαριστώ κύριο Σάλβαρο. Ζήτησε το λόγο και μετά θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να απαντήσει στο θέμα το αριθμητικό που έθεσε ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Τι άλλο να προσθέσει ο εισηγητής σχετικά με τις τρεις αυτές περιπτώσεις. Δεν θέλω να προκαταλάβω βέβαια. Τέλη Απριλίου θα ασχοληθεί η Επιτροπή με το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Αυτά που είδαμε πέρσι ήταν ένα πρώτο κύμα. Τώρα από τη Γερμανία μπορώ να σας αναφέρω μια λίστα τουλάχιστον 20 μικρών και μεσών επιχειρήσεων όπου θα ζητήσουν υποστήριξη από το Ταμείο αυτό και αφού η Κομισιόν είναι παρούσα. Μήπως μπορεί να μας εξηγήσει πώς θα λειτουργήσει το θέμα στο μέλλον εν και του μηδενικού περιθωρίου που διαθέτουμε. Και δεν υπάρχει από πουθενά να βρούμε χρήματα. Πώς θα υλοποιηθούν αυτά στο μέλλον. Διότι η αξίωση δεν είναι δεδομένη, αντίθετα από ότι για την κοινή αγροτική πολιτική. Αν μπορεί να κάνει κάποια σχετική εκτίμηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι θαυμάσιο για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια ερώτηση προς τον εισηγητή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δεύτερο δοσιά της Λιθουανίας. Μιλούμε για κάποιες οικοδομικές εργασίες. Το ταμείο αυτό είναι ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Άρα προορίζεται μάλλον για τη βιομηχανία που έχει θυγεί από το ανταγωνισμό άλλων χωρών. οικοδομικές δραστηριότητες στις μικρές ε, οικοδομικές επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει αυτός ο στιγνός ανταγωνισμός από τις άλλες ε, χώρες. Σίγουρα θέλουμε να βοηθήσουμε βέβαια τη Λιθουανία για να εξέλθει από την κρίση. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης ε, ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο πρόβλημα του οικοδομικού κλάδου της Λιθουανίας. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαντήσει, ή να κάνει κάποια σχόλια. Ο Γενικός Διευθυντής και μετά ο κύριος Μπέγκε. Ευχαριστώ. Θα σας δώσω κάποιες εξηγήσει και μετά θα δώσω το λόγο στην συνάδελφα από τη Γενική Διάθεση Απασχόλησης για άλλα σημεία. Σε ό,τι αφορά το αίτημα της Λιθουανίας και την προθεσμία. για τη συμπερίληψη του αιτήματος αυτού που υπευλήθη 23 Εβδόμου. Πολύ πριν δηλαδή το πρώτο αίτημα της επιχείρησης Κάρμαν και το δεύτερο αίτημα την αίτηση που υπευλήθη στις 23 Ενάτου 2008. Η απάντηση είναι απλούστατη. Υπήρχαν, υπήρξαν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που χρειάστηκε για να προωθηθεί το δοσιέ και αυτές οι τεχνικές ε, λεπτομέρειες ζητήθηκαν από την λιθουανική κυβέρνηση. Αλλά επειδή μεσολαβούσαν οι θερινές διακοπές, τις απαντήσεις λάβαμε εκπρόθεσμα. Γι' αυτό δεν προλάβαμε να δρομολογήσουμε αυτό το ντοσιέ, γιατί μας έλειπαν στοιχεία. Ήταν ε, ατελές το σχέδιο της Λιθουανίας. Σε ό,τι αφορά τα ποσά, θα το διευκρινίσει και συνάδελφος. Το θέμα αυτό το έχουμε ήδη ξανασυζητήσει. Δηλαδή υπάρχει διαφορά μεταξύ του αριθμού των εργαζομένων που εθίγησαν άμεσα από το μέτρο της απόλυσης που απολύθηκαν δηλαδή εξαιτία της οικονομικής κρίσης και των εργαζομένων που δίνανται να επωφεληθούν από την συνδρομή αυτή, από την βοήθεια αυτή, αν και ορισμένοι από αυτούς ήδη έχουν ξαναβρει μια δουλειά και άρα δεν χρειάζονται αυτή τη συνδρομή. Ίσως όμως θα μπορούσε να σας διαφωτίσει καλύτερα εδώ η συνάδελφος από την ε, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν θέλετε κύριε Πρόεδρε μπορούμε να της δώσουμε το λόγο. Όπως ξέρετε, τα κράτη-μέλη έχουν 10 εβδομάδες στη διάθεσή τους μετά την περίοδο αναφοράς προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους. Και μέσα σε αυτές τις 10 εβδομάδες συγκεντρώνουν τα στοιχεία και βλέπουν πόσοι καλύπτονται από τα μέτρα αυτά. Στο μέτρο που τα κράτη-μέλη αποκτούν πείρα με τη χρήση του Ταμείου παγκοσμιοποίηση. διαπιστώνω ότι δεν χρειάζεται να βάλουν στον προπολογισμό το μέγιστο αριθμό δικαιούχων. Καλύτερα να εστιάσουν τα μέτρα σε εργαζόμενους που πραγματικά θέλουν να, ε, να τα εφαρμόσουν. Οπότε έχουν πολύ πιο γρήγορα επαφές με τους εργάτες, ε, ε, κάνουν τα σχέδιά τους γιατί μέτρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν και ασχολούνται με τους πραγματικά ενδιαφερόμενους εργάτες. Οι εργάτες στόχος είναι αυτοί που ήδη εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι ίσως έχουν στο μεταξύ βρει άλλη δουλειά ή ίσως έχουν αποφασίσει να συνταξιδοτηθούν. Οπότε δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμπερίληψη στα μέτρα. Με ρωτήσατε πόσες αιτήσει περιμένουμε για τους επόμενους μήνες. Τα κράτη-μέλη έχουν διάφορες ε, περιπτώσεις. Έχουμε ήδη διαβουλεύσεις. Τώρα, πόσες από αυτές θα καταλήξουν σε επίσημες αιτήσει δεν ξέρουμε. Θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των κρατών μελών. Πάντως, πέρυσι λάβαμε 29 αιτήσει και μέχρι στιγμής ε, ούτε οι μισές δεν έχουν φτάσει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Ήδη προωθούμε τις αιτήσει ε, που ήδη λάβαμε, αλλά και περιμένουμε νέες αιτήσει. Σε ό,τι αφορά τον οικοδομικό κλάδο, τον κατασκευαστικό κλάδο, όντως δεν πρόκειται για ένα κλάδο που ε, πλήγεται άμεσα από την παγκοσμιοποίηση που συνδέεται με το εμπόριο. Πάντως μετά την περσινή αναθεώρηση του κανονισμού, προβλέπετε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, που από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους, έτσι λέει ο κανονισμός, οι εργαζόμενοι που ε, θίγησαν άμεσα από τις απολύσεις που σχετίζονται με την παγκόσμια οικονομική κρίση μπορεί να περιληφθούν στον κανονισμό όπως οι, εργαζόμενοι που απολύθηκαν εξαιτίας ε, των εμπορικών συνεπειών της παγκοσμιοποίησης. Ο εισηγητή δεν έχει άλλε παρατηρήσει. Την άλλωστε η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό άλλη φορά με τι διευκρινήσει που ζητήσαμε. Αν δεν θέλει άλλο κανεί το λόγο, σα ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρίαση. Ραντεβού αύριο στι 9. Σα θέλω παρακαλώ να είστε συνεπεί αύριο και στην ώρα σα στι 9 γιατί έχουμε ψηφοφορίες και απαιτείται απαρτία. Θα ήθελα όμως να παραμείνουν στην αίθουσα οι συντονιστές. και οι εισηγητές των προπολογισμών 2010 και 2011, αλλά κυρίως 2010, κυρίως ε, εσάς εννοώ κύριε Μάνικα, γιατί έχουμε ένα απροσδόκητο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Και όποιοι από το Προεδρείο μπορούν να παραμείνουν ε, είναι ευπρόσδεκτοι.